Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να σας καλωσορίσω όλους. Ξεκινάμε λοιπόν με την έγκριση των, της ημερήσιας διάταξης και να σας υπενθυμίσω ότι γίνεται web streaming της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ να είμαστε προσεκτικοί στα όσα λέμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο σημείο που είναι η έγκριση της ημερήσιας αδιάταξης. Ο κύριος Ντεάντζελης, ο οποίος πρέπει να φύγει, έχει νωρίς αεροπλάνο. Έχει μία γνωμοδότηση έχει μια γνωμοδότηση αύριο στο σημείο 17. Θα τη μεταφέρουμε στη σημερινή ε, απογευματινή συνεδρίαση και θα τη συζητήσουμε μετά το σημείο 13. Εάν δεν υπάρχει καμία παρατήρηση, θεωρώ πως έχει εγκριθεί το πρόγραμμα της της διάταξης. Περνάμε στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών της 6ης Σεπτεμβρίου και της 27ης και 28ης Σεπτεμβρίου. Έχουν μοιραστεί και στο τέλος της συνεδρίας θα θεωρήσουμε πώ έχουν εγκριθεί, αν εντωμεταξύ δεν ακουστούν ενστάσεις. Παρακαλώ πολύ. Η συνάδελφος μας ανακοινώσατε πως το 17 θα το συζητήσουμε μετά το 13. Όμως για μένα αυτό σημαίνει πως το δικό μου αναβάλλεται για αύριο το απόγευμα. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Σας ευχαριστώ πάντως Κωνσταντσα που α, μίλησες ελεύθερα για αυτή την ανησυχία σου. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3. Εδώ έχω δύο ανακοινώσει που θα ήθελα να κάνω. Καταρχήν να σας πενθυμίσω όταν εάν πηγαίνετε στη Ρουμανία πως το ταξίδι αυτό θα γίνει 3 με 5 Νοεμβρίου και πως το ταξίδι αυτό Στο ταξίδι αυτό συμμετέχουν 11 μέλη της Επιτροπής μας, 5 είναι Ρουμάνοι. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, επιτόπου και κυρίως στις περιοχές της Μοσοάρα, Άράτ και Τζούτζου. Θα συναντηθούμε εκεί με τους τοπικούς ε, πολιτικούς ε, άτομα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Φανλίστερο είναι, ε, έχει την προεδρία αυτής της αποστολής και για όσους θέλουν παραπάνω προφορές για αυτή την αντιπροσωπεία μπορείτε να πάτε στο website μας ε, και να βρείτε τις προφορίες είτε να απευθυνθείτε κατευθείαν απευθείας μάλλον στη γραμματεία. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω πως την περασμένη εβδομάδα στις 19 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, στο Στρασβούργο, η Επιτροπή ε, ενέκρινε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο έχουμε ένα σημαντικό τμήμα που ε, αναφέρεται στην πολιτική συνοχή. Για όσους δεν το έχουν ε, και δεν έχουν εξοικειωθεί με τα όσα συμπεριλαμβάνονται, να σας πω πως το έγγραφο αυτό είναι διαθέσιμο και μπορούμε να το δούμε όλοι. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Για πρώτη φορά Έχουμε εκπρόσωπο εδώ από ένα κράτος μέλος, έχουμε τον Υπουργό Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας, έχουμε τον κύριο Ρόζεν Πλευνέλιεφ μαζί μας και είμαστε ευγνώμονες και πιστεύω ότι εκφράζω όλη την Επιτροπή για την τιμή που μας κάνετε και ελπίζω πως όλοι οι συνάδελφοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για την κατάσταση ε, στην Βουλγαρία και στα πλαίσια της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, με αλλά και στα πλαίσια της εφαρμογής ε, των πολιτικών για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 και χαίρομαι για μια φορά ακόμη και σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση. Θα σας δώσω το λόγο και μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Θα γίνει μια εισαγωγή και μετά μπορούμε να συζητήσουμε κάποια θέματα και να σας επευθύνουμε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που μας δίνετε την ευκαιρία να σας απευθύνουμε τον λόγο για το που βρίσκεται η Βουλγαρία τώρα και προς τα που κατευθύνεται η πολιτική συνοχής και η εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων στην Βουλγαρία. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Είμαι πρόσφατα έγινα υπουργό πριν από ένα χρόνο και λίγο περισσότερο και για τα δημόσια έργα και είμαι υπεύθυνο για δύο από τα 7 βουλγαρικά λειτουργικά προγράμματα με κάθε σεβασμό που έχω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας βεβαιώνω ότι βελτιώνουμε και την επικοινωνία και την συνεργασία και την απόδοσή μας και μπορούμε να το αποδείξουμε. Στο <clears throat> Υπουργείο μας αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και αποφασιστικά και κάνουμε αποφασιστικά βήματα για να εξασφαλίσουμε διαφάνεια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων στους τομείς όπου είμαστε υπεύθυνοι εμείς και το Υπουργείο μου δηλαδή. Έχουμε κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις βέβαια, έχουμε προβλήματα και βέβαια έχουμε σημειώσει καθυστερήσεις, έχουμε όμως μια στρατηγική, έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό και προχωρούμε. Τι έχουμε κάνει λοιπόν. Πρώτα βελτιστοποίησαμε το σύστημα ε, καταβολών προς τους ε, απολύπτες με ε, ένα σύστημα για πιο εύκαμπτη διαχείριση των ταμείων και κάνουμε και δειγματοληπτικούς ελέγχους επιτόπου. Έχουμε μειώσει τον χρόνο για την επαλήθευση των αξιώσεων και κάνουμε και εκ των προτέρων έλεγχο των εγγράφων των ε, εποφελουμένων, των απολυπτών και στις ε, διάφορες διαδικασίες πρόσκληση ενδιαφέροντος κτλ. Επίσης ρίχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην διαφάνεια. Κάνουμε, έχουμε ε, βελτιώσει και έχουμε ε, ενημερώσει τις ε, σχέσεις με τους απολύπτες. Τα συνδιαδημοσιεύουμε και στο διαδίκτυο dgregio.eu για όλες αυτές τις εφαρμογές. Έχουμε κάνει και ημερίδες ενημέρωσης και στο περιφερειακό επίπεδο αλλά και στο τοπικό επίπεδο. Για κάθε δημόσιο πρόγραμμα έχουμε βελτιώσει την μεθοδολογία για την επαλήθευση και ρύθμιση των τιμών. Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε συστήσει και επιτροπές που είναι απαραίτητες και έχουμε βάλει και εφόσον χρειάζεται αυτό και εξωτερικούς ε, αξιολογητές από διαφορετικούς οργανισμούς, ιδίως από το Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων, το Εμπορικό Επιμελητήριο και το Επιμελητήριο των Σχεδιαστών επίσης ε, του Βουλγαρικού Επιμελητηρίου Οικοδομικών Επιχειρήσεων, από το εξωτερικό επίσης κλπ. Έχουμε περιλάβει επίσης μεταξύ αυτών των εμπειρογνωμόνων ομάδες οι οποίες συμμετέχουν ως αξιολογητές σε όλα τα προγράμματα δημοσίων προμηθειών και ειδικού εκπροσώπους από τις οργανώσεις των αναπήρων στην Βουλγαρία. Αρχίσαμε επίσης μια νέα πρωτοβουλία κατά της διαφθοράς για το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα. Έχουμε βάλει και την Transparency International να συμμετέχει ως ε, εποπτική αρχή. Έχουμε δημοσιεύσει και δημοσιεύουμε ε, στο διαδίκτυο όλα τα μεγάλα έργα έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν από την αρχή, να μην ευνηδιάζονται δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι και να μπορούν να κάνουν τα σχόλια τα οποία εμείς μετά προσέχουμε ιδιαίτερα. Πού βρισκόμαστε τώρα. 30 ε, προγράμματα έχουν ξεκινήσει τώρα με 23 δισεκατομμύρια ή 77% του επιχειρησιακού προγράμματος. Ο αριθμός είναι συνολικά 1895 με συνολικό, το συνολικό ποσό, και αυτά είναι ξεκάθαρα νούμερα, είναι 67 εκατομμύρια. Σημαντική είναι και η επιτυχία μας στην αύξηση της ταχύτητας για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών το 2007 δεν καταφέραμε να κάνουμε πολύ χαμηλή απορροφητικότητα, το αντιμετωπίζουν όμω και άλλε χώρε αυτές. Αυξήθηκε σημαντικά το 2008, 254.000 το 2009 και 304 εκατομμύρια το 2010. Ε, Αυτό δείχνει καθαρά ότι το 2010 έχουμε φτάσει στο 2,5 φορές, 2,5 φορές από το 2008. Και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 53% του προπολογισμού του OPRD μέχρι το τέλος του 2010. Έχουμε και στόχο για το 2011 που φτάνει το 90% ανάθεση. Το συνολικό ποσό βέβαια εξακολουθεί να παραμένει το μέγα πρόβλημα. Αλλά και πάλι τα γεγονότα τώρα ποια είναι. Το 2007 αυτά που καταβάλαμε ήταν 0. Το 2008 2 εκατομμύρια ευρώ. Το 2009 28 εκατομμύρια ευρώ και το 2010 έχουμε περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ. Η καταβολή λοιπόν των πόρων έχει αυξηθεί σημαντικά. Έξι φορές ταχύτερα από το 2009 μέχρι το 2010. Βέβαια ήταν χαμηλές ε, αρχικά οι καταβολές. εντιμετωπίζαμε προβλήματα, αλλά ποια είναι τα γεγονότα. Ήδη έχουμε φτάσει 70% πληρωμών από το συνολικά, από το συνολικά ανατεθειμένο ποσό. Συνοψίζοντας λοιπόν, το, η ταχύτητά μας αυξάνεται σημαντικά. Έχουμε φτάσει και σε υψηλότερο ποσοστό από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και ελπίζουμε στο μέλλον να καταφέρουμε να γίνουμε από τους πιο αποδοτικούς. Τώρα, επίσης σημαντικό, οι βουλγαρικές τοπικές κοινότητες έχουν βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητά του τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, πλήγηκαν σοβαρά από την κρίση. Οι προπολογισμοί τους μειώθηκαν σημαντικά πράγματι. Και τα ευρωπαϊκά ταμεία όντω είναι η μοναδική σωτηρία για πολλέ από αυτέ τι κοινότητε. Πιθανώς όμως λόγω της κρίσης και λόγω του σωστού χρονισμού μπόρεσαν να ρίξουν ιδιαίτερη προσοχή ε, σε ορισμένα προγράμματα και τα τελευταία 1,5 χρόνια βλέπουμε στον αγωγό να είναι όριμα πλέον ε, κοινοτικά έργα τα οποία δεν ήταν καθόλου έτσι πριν από 1,5 χρόνο. Έχουμε λοιπόν μια στέρεα βάση και αυτό είναι σαφές ότι το λειτουργικό μας πρόγραμμα για την περιφερειακή ανάπτυξη θα έχει μια λίστα αναμονής καλών έργων και πολύ πριν από το 2014 θα έχουμε ευθυγραμμιστεί ώστε να αποδίδουμε καλά και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Και μιλώντας για το μέλλον, πρέπει να πούμε κάτι σαφώς, ότι το Υπουργείο μας συμμετέχει ήδη στις συζητήσεις. Το Υπουργείο μας καθορίζει τους νέους στόχους της πολιτικής συνοχής για τις βουλγαρικές προτεραιότητες. Εργαζόμαστε πραγματικά από τις ρίζες προς τα πάνω με διαφορετικά εργαλεία και μέσα διοικητικά και άλλα, για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Ήδη το Υπουργείο μας έχει αρχίσει τον προγραμματισμό για το 2014 έως 2020. Έχουμε ήδη αρχίσει να μελετάμε τους στόχους της ε, περιφερειακής συνοχής και δίνουμε και προτεραιότητα σε ε, τομείς προβληματισμού και στις ειδικέ επενδύσεις. Και βέβαια λόγω της αρνητικής, των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης οι τοπικές αρχές έχουν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα για το μέλλον. Είναι απαραίτητο η πολιτική συνοχή να αντιμετωπίσει τις βασικές ανάγκες των αρχών αυτών. Χρειάζεται λοιπόν ε, μέσα δικότητα της ενέργειας, χρειάζονται δρόμους, χρειάζονται αποχετευτικά έργα, χρειάζονται υδροδότηση, χρειάζονται επένδυση σε υποδομές και οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι αυτές οι βασικές ανάγκες της υποδομής δεν είναι μια απλή ανάγκη, ούτε είναι πολυτέλεια, ούτε κάτι που δεν και καλά θέλουμε. Αυτό που χρειάζονται οι περιφέρειές μας, ε, οι πόλεις μας, ο βουλγαρικός βοράς που είναι και από τις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης χρειάζεται να αναπτυχθεί. Και για να αναπτυχθεί βασικό μέσον είναι οι υποδομές. Χρειάζεται λοιπόν να προλάβουμε του υπολείπου. χρειάζεται να αναπτυχθούμε και για το λόγο αυτό χρειάζεται να γνωρίζουμε τι να περιμένουμε από την πολιτική συνοχή η οποία απευθύνεται σε αυτούς τους τομείς ακριβώς. Επίσης ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δημιουργεί πολλά προβλήματα για την ώρα στην βουλγαρική κυβέρνηση το πρόγραμμα των μεταφορών. Εγώ είμαι υπεύθυνο για τους δρόμους, επειδή είμαι και υπεύθυνο για τα δημόσια έργα. Γνωρίζουμε ότι ορισμένα από τα πιο σημαντικά έργα βρίσκονται σε καθυστέρηση και μας ανησυχεί αυτό. Αλλά έχουμε ένα σχεδιασμό και έχουμε σκοτωθεί στη δουλειά. Και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο το οποίο ελέγχεται έχουμε μια ειδική μονάδα συντονισμού και ένα πρώτο πρόγραμμα οδικής υποδρομής 150 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου ήδη έχει ξεκινήσει για 250 εκατομμύρια ευρώ και αναμένουμε ολοκλήρωση το 2012. Αυτός ο αυτοκινητόδρομος θα είναι και ένα μέρος των, ε, των ε, διαδρόμων 4 και 8, των Ευρωπαϊκών Διαδρόμων 4 και 8. Και πάλι εκεί μας ελέγχει η Transparency International. Τους επόμενους 6 μήνες, θα σας λέω καθαρά, ότι θα είναι σημαντική για μας, κρίσιμη για μας για τις μεταφορές μας. Χρειάζεται να προχωρήσουμε ταχύτερα με το OP Transport. Χρειαζόμαστε νέες προσκλήσεις εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και να αυξήσουμε τη διοικητική μας ικανότητα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να εφαρμόσουμε. Και εδώ όμως έχουμε ξεκάθαρους στόχους, οι οποίοι είναι ότι μέχρι τέλη του 2010 θα φτάσουμε στο 25% ανατεθειμένων έργων και μέχρι το 2011 66% και μέχρι το 2012 100%. Και οι στόχοι μας για την εφαρμογή, βρισκόμαστε βέβαια πολύ χαμηλά τώρα, μόλις 4%, αλλά θέλουμε 23% να φτάσουμε μέχρι το τέλος του 2011 και να φτάσουμε 50% μέχρι τα τέλη του 2012 συζητήσαμε και το θέμα του overbooking. Έχουμε 40% overbooking για την τρέχουσα περίοδο, κάτι το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Εντοπίσαμε όμως όχι μόνο την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το overbooking, αλλά και συγκεκριμένα έργα και αυτά εντάσσονται μέσα στις βουλγαρικές εθνικές προτεραιότητες και μέχρι το 2020 και επιζητούμε την υποστήριξη των διεθνών IFI για τα ε, έργα εκείνα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας και τα οποία θα ενταχθούν στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού που γνωρίζουμε ότι έχουμε μονάχα τρία χρόνια για να προετοιμάσουμε τα έργα αυτά και γνωρίζουμε ότι πρέπει να αναλυθεί ταχαίως δράση. Έχουμε κάνει τις σχετικές αιτήσει και βέβαια είμαστε ανοιχτοί στον συντονισμό και στη συνεργασία με τους IFI για να επιταχύνουμε την διαδικασία αυτή. Και βέβαια χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Βουλγαρία συμμετέχει ήδη στην προσπάθεια της αναθεώρησης των ε, διευρωπαϊκών δικτύων με προτάσεις και έχουμε έναν αυτοκινητόδρομο που είναι και που ε, ενώνει όλα τα Δυτικά Βαλκάνια και ε, θα επιζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη για να μπει ο αυτοκινητόδρομος αυτός στα αναθεωρημένα διευρωπαϊκά δίκτυα και για τη στατική του Δούναβη τώρα, επειδή είμαι και εθνικό συντονιστή για την στατική του Δούναβη, σίγουρα θα ε, τεθούν ερωτήσεις και για το θέμα αυτό. Η Βουλγαρία υποστηρίζει την ιδέα αυτή. Εμείς είμαστε υπερήφανοι που για την ε, στατική και πολιτική του Δούναβη έχουμε ξεκινήσει από τα κάτω, ε, από τις ρίζες, με τους δημάρχους, τους κοινοτάρχες, με τα πανεπιστήμια του Βουλγαρικού Βορρά Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζουμε το σχέδιο δράσης και αναμένουμε βέβαια με μεγάλη ανυπομονησία την έγκριση του σχέδιου δράσεως. Επίσης, θέλουμε να ενταχθούμε και εμείς στρατηγική αυτή τη ε, διαπραγματεύσεως της νέας ε, ε, δημοσιονομικής προοπτικής. Με το σωστό σχεδιασμό η βουλγαρική κυβέρνηση ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες αυτές και έχουμε αρκετό χρόνο για να τις θέσουμε σε εφαρμογή. Βέβαια, είμαστε ευγνώμονες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ιδέα της στρατηγικής του Δουναβή, η οποία μας επιτρέψει να παραγάγουμε ε, έργα που είναι διαπεριφερειακής σημασίας για, την, ε, για, για μεγάλα ε, έργα ναυαρχίδες, flagship projects δηλαδή, Έχουμε, ένα, έχουμε δύο μεγάλα έργα τα οποία βρίσκονται το ένα στη φάση σχεδιασμού και το άλλο στη φάση της κατασκευής και χρειαζόμαστε βέβαια να συνθέσουμε τις ε, χώρες του Δούναβη. Η Βουλγαρία λοιπόν είναι διατεθειμένη και να συμμετάσχει και να αναλάβει ηγετικό ρόλο, να προωθήσει όλες ε, τις μορφές συνεργασίας και πολιτιστικής και τουρισμού, γιατί αυτό αποτελεί προτεραιότητα για τη βουλγαρική κυβέρνηση, μαζί βέβαια με τη Σερβία καθώς και άλλες γειτονικέ χώρες, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινό έργο, μια νέα στρατηγική δηλαδή, του Δούναβη, που θα συνδέσει και τουριστικούς ε, τόπους και θα δώσει και την πολιτιστική διάσταση. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο. Προσπάθησα μέσα στο σύντομο χρόνο να αναφερθώ σε πολλά θέματα και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε αλλά και με τις προσπάθειες που κάνει η βουλγαρική κυβέρνηση. Και σας ευχαριστώ πολύ που σε αυτή την περίοδο ειλικρίνειας και ανοιχτού διαλόγου δεχτήκατε να έρθετε ε, εδώ και να μας κάνετε αυτή την παρουσίαση και θα ήθελα να δώσω και στην Υφυπουργό το λόγο και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε είτε με ερωτήσεις ή μάλλον πρώτα απ' όλα ε, ερωτήσεις και μετά θα ακούσουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Μποστινάρου, ο οποίος όμως θα το δώσει στην συντονίστρια του και αυτός με τη σειρά του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι πολύ που μας φέρνετε θετικά νέα από την Βουλγαρία, γιατί οι πληροφορίες που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες εδώ στις Βρυξέλλες δεν ήταν τόσο θετικά και μας ανησυχούσαν πολύ σχετικά με το ότι η Βουλγαρία αλλά εν μέρη και η Ρουμανία δεν είναι η θέση να απορροφήσουν τους μεγάλους πόρους που θέτει στη διάθεσή τους η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε καταβάλουν τις σχετικές προσπάθειες. Λυπούν πολύ, ειδικά σήμερα το πρωί έλαβα από τον κύριο Κοντμάνης της φιλελεύθερης ομάδας που είναι και εισηγητής για την Επιτροπή Προϋπολογισμών για την πολιτική συνοχή ιδιαίτερα έλαβα ένα έγγραφο που λέει ότι η απορρόφηση και οι πραγματικές πληρωμές στον τομέα της πολιτικής συνοχής βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν έχουν αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο ας πούμε. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Γνωρίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ότι οι πόροι για την βελτίωση της διοίκησης απορροφώνται σωστά, από την άλλη μεριά οι διοικήσεις δεν λειτουργούν καλά, διότι πολλοί από τους εκπαιδευμένους υπαλλήλους αμέσως μετά από την εκπαίδευση αυτή αφήνουν τη δημόσια διοίκηση και προσλαμβάνονται σε ιδιωτικέ επιχειρήσει. Εν πάση περιπτώσει δεν βρίσκονται πλέον στην διάθεση των δημοσίων διοικήσεων που ε, υποτίθεται ότι θα ε, προωθήσουν τα έργα αυτά στην Βουλγαρία. Πού οφείλεται αυτό, έχετε κάποια ιδέα, έχετε επίση κάποια ιδέα πώ μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση στην χώρα σα διότι ο στόχο και βέβαια θέλουμε την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο πρώτος στόχος της διοικητικής αρρωγής είναι να βελτιωθούν οι αποδόσεις των διοικήσεων, ώστε να μπορούν μετά με τη σειρά τους να συμβάλλουν στην ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων. Δεύτερη ερώτηση, επειδή μου ετέθη υπόψη το θέμα, επειδή με συντονίστηκε της πολιτικής μου πριν από λίγο καιρό κατατέθηκε μια αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα μεγάλο έργο για την ανακύκλωση αποβλήτων στη Σόφια, είναι γεγονός ότι όντως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καθόλου αυτό και ότι τα απορρίμματα εξακολουθούν να μεταφέρονται εκατοντάδες χιλιόμετρα διαμέσου της Βουλγαρίας για να καταλήξουν κάπου αλλού. Πού βρίσκεται το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να μιλήσω τη γλώσσα μου. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθατε στη δική μας Επιτροπή για να συζητήσουμε τα θέματα της περιφερειακής πολιτικής. Να ξαναμιλήσω όμως αγγλικά, αφού σας καλωσόρισα στα βουλγαρικά. Λοιπόν, πείτε μου, το προσωπικό το οποίο απασχολείται στην υπηρεσία, υπηρεσία ε, σιδηροδρομικού υλικού και εξοπλισμών μειώθηκε κατά 50% στην αρχή της χρονιάς. Και πείτε μου, είναι στην περιοχή Στράσπροτ όπου η καθυστερήση στην απορρόφηση κονδυλίων είναι η μεγαλύτερη και όπου ελοχεύει ο κίνδυνος τα κονδύλια αυτά να χαθούν. Τι μέτρα θα πάρετε για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση, αν όντω είναι έτσι. Δεύτερον, την επόμενη επιτροπή, η Επιτροπή Ρέτζι, θα πάει στη Ρουμανία. Όμως η δική μου πρόταση και οι συνάδελφοι από τους, φιλοδελ... την... Ε, μας είχαν πει πω θα πρέπει να πάμε στη Βουλγαρία στο Τζούρτζου. Στο Τζούρτζου λοιπόν αυτό που είχαμε σκοπό να συζητήσουμε ήταν τη διασυνοριακή συνεργασία στα πλαίσια τη στρατηγική για το Δούναβη. Και εδώ σα ερωτώ κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα μεγάλα έργα μέσω των οποίων η Βουλγαρία προβλέπει να δώσει σάρκα και οστά στη συνεργασία με τη Ρουμανία και ενδεχομένω όχι μόνο με τη Ρουμανία αλλά και με άλλους για να δρέψει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η στραγική για, την, ε, για το Δουναβική με το δήμαρχο του Ρούσε, τον οποίο εμείς στο Τζούτζου θα συναντήσουμε. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να του στείλετε για τη διασυνοριακή συνεργασία με τη Ρουμανία. Και πείτε μου, μια επιπλέον ερώτηση, πώς αξιολογείτε εσείς τη συνεργασία και την εταιρική σχέση με τους εταίρους μας από τη Ρουμανία τη στιγμή του σχεδιασμού και την εφαρμογή της στρατηγικής για το Δούναβη. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε ε, στις επόμενες ερωτήσεις να σας υπενθυμίσω πως έχουμε επισκέπτες από τις Ηνωμένε Πολιτείες είναι λοιπόν εκπρόσωποι μεγάλων αμερικανικών εταιριών που έχουν έρθει εδώ στις Βρυξέλλες να βρουν ευκαιρίες επιχειρηματικές. Και χαίρομαι που είστε εδώ, σας καλωσορίζω. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα. And now, uh, Κυρία Χιουσμένοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την ε, παρουσία σας εδώ σήμερα και για τα όσα μας είπατε ε, τώρα το απόγευμα. Τις επόμενες ημέρες, μάλλον αύριο και σήμερα το απόγευμα, θα μιλήσουμε για τις προτεραιότητες για την πολιτική συνοχή. Και νομίζω πως τα συμπεράσματα που έχουμε μπροστά μας και τα, τα στοιχεία που έχουμε θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βάση για να συνάγουμε κάποια συμπεράσματα διαφορετικά λίγο από αυτά που αναμέναμε. Βλέπουμε από τα όσα μας είπε ο Υπουργό πως η πολιτική συνοχή λειτουργεί. Αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα το οποίο μπορεί να ε, εξάγει κανείς από ένα κράτος το οποίο πολύ πρόσφατα έγινε μέλος και που είναι μάλλον η μοναδική του επιτυχία. Ξέρουμε πώς είναι τα προβλήματα ε, και ποιε είναι οι προκλήσεις για τη συνοχή. Καταρχήν έχουμε τον χαμηλό ρυθμό απορρόφησης. Αλλά αυτό το ε, συμβαίνει και σε άλλα κράτη. Ίσως λοιπόν ε, θα έπρεπε να μετράμε την ποιοτική ε, διάσταση, όχι τόσο την ποσοτική. Τώρα για την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν αυτά τα project, να σας πω ποιος είναι ένας από τους στόχους της Βουλγαρίας. Να έχουμε ορατά αυτά αποτελέσματα τα οποία να αναγνωρίσουν οι συμπολίτες μας. Και πιστεύω πως η πολιτική συνοχή θα πρέπει να μετρηθεί με γνώμονα την ε, προστιθέμενη αξία που προσφέρει. Σας ευχαριστώ. για το ότι η στρατηγική για το Δούναβι είναι πλέον προτεραιότητα για την ε, βουλγαρική κυβέρνηση και νομίζω ότι σε επίπεδο συζήτησης για το θέμα αυτό υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ των ε, μικρών των κυβερνητικών φορέων και των ε, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. ρωτώ όμως το εξής. Η κυβερνητική στρατηγική αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα σκαριά και δεν ξέρω αν ε, σκέπτεται να κατασκευαστεί και μια τρίτη γέφυρα γιατί νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί κάτοικοι του Δούναβη που θα πετούσαν τις περιοχές γύρω από το Δούναβη που θα πετούσαν κάτι τέτοιο. Μπορείτε εσείς να πείσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλετε και μια τρίτη γέφυρα. Λοιπόν, μπορείτε να αποφασίσετε σε αυτά τα σχόλια και μετά θα ακούσουμε τους επόμενους συναδέλφους. Ο Υπουργός στα Γερμανικά. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις ήταν πολύ σημαντικές και με την ευκαιρία θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ευθύς αμέσως. Έχουμε τα συγκεκριμένα γεγονότα τώρα. Είπατε βέβαια και σωστά η βουλγαρική εικόνα, αυτό το image, εξακολουθεί να είναι ευάλωτο, ας το πούμε, ευάλωτη εικόνα βρίσκομαι ενώπιόν σας, αλλά οι ειδήσει από τη Βουλγαρία δεν είναι τόσο θετικές. Εδώ υπάρχουν δύο ξεκάθαρα πράγματα που μπορώ να σας πω. Και εγώ διαβάζω καμιά φορά ε, τις ειδήσει και μου φαίνεται ότι η καλύτερη ειδήση είναι η χειρότερη. Ε, αλλά ποια είναι τα γεγονότα. Τώρα, ε, η γεγονό είναι ότι τα πρώτα μεγάλα έργα αρχίζουν ήδη να κατασκευάζονται. Για παράδειγμα, ο αυτοκινητόδρομος που ανέφερα, που αποτελεί τμήμα δύο ευρωπαϊκών διαδρόμων, με 300 εκατομμύρια ευρώ, άλλος με 250. Είναι σαφές ότι ήμασταν το προβληματικό παιδί και εξακολουθούμε να είμαστε. Αλλά δουλεύουμε σκληρά. Έχουμε έναν σχεδιασμό, έχουμε χρονοδιαγράμματα, έχουμε πολύ ξεκάθαρη στόχευση και έχουμε εντελώς αποπολιτικοποιήσει τις δομές αυτές. Μας ενδιαφέρουν μονάχα τα αποτελέσματα στο επίπεδο των εμπειρογνωμόνων και γι' αυτό ελπίζουμε τους επόμενους έξι μήνες να ξεκινήσουμε άλλα 7 μεγάλα έργα. Έχετε λοιπόν απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι πάνω από 1,2 εκατομμύρια Βούλγαροι έχουν φύγει στο εξωτερικό και είναι άνθρωποι εκπαιδευμένοι με προσόντα. Αλλά στην περιφερειακή ανάπτυξη το τμήμα που έχουμε για να παρακολουθεί αυτήν έχει 166 άτομα προσωπικό. Όλοι νέοι και όλοι με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Όπως είδαμε με τα γεγονότα, έχει, έχει τριπλασιαστεί η ανάθεση έργων για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν καινούριου μηχανισμούς μπόνους. Ε, έχουμε το μηχανισμό διπλού εισοδήματος όπως τον αποκαλούμε και ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Τα σημάδια ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο είναι ε, πραγματικά και για άλλους οργανισμούς που έχουν σχέση με τα ευρωπαϊκά ταμεία οργανισμός δηλαδή οδών. Μιλούμε τώρα εκεί, σχεδιάζουμε τώρα ένα τελείω τελείως διαφορετικό κόνσεπτ για τις πληρωμές. Γιατί η κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόμου διαρκεί 3-4 χρόνια και οι άνθρωποι πρέπει να ε, διαθέτουν τη δέσμευση και τον ενθουσιασμό για να εργαστούν όλο το διάστημα αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα payment and motivation scheme για τους αυτοκινητοδρόμους. Και μια τελευταία φράση. Η Όλαφ επιβεβαίωσε ότι η Βουλγαρία είναι τώρα πολύ διαφανέστερη και ότι έχει βελτιωθεί πολύ και η επικοινωνία. Τώρα τα απορρίμματα στη Σόφια. Όλοι ανησυχούμε για το έργο αυτό και για την μεταφορά των απορριμμάτων. Όμως τώρα έχει ληφθεί η απόφαση για το έργο, θα υπάρξουν διάφορες φάσεις και οι εμπειρογνώμονες δουλεύουν νυχθημερών μαζί με τους εταίρους μας και τους συνεργάτες μας εδώ στις Βρυξέλλες. Θα βρεθεί η λύση. Η Σόφια βέβαια έχει ακόμα το πρόβλημα αυτό, το οποίο βεβαίως πρέπει να λυθεί το δυνατόν σύντομότερο. Υπάρχει πάντως ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Μέχρι τέλους του έτους θα έχει ε, ολοκληρωθεί κατά 100%. Να σας πω λοιπόν για τον οργανισμό σιδηροδρόμων πως όντως οι πληροφορίες που έχετε είναι σωστές και βεβαίως ε, χαίρομαι που είναι τόσο ενημερωμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Είχαμε απολύσεις εκεί όντως. Δεν ήταν το 50% του προσωπικού αλλά ήταν ένα μεγάλο κομμάτι και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω Αυτή τη στιγμή έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς, για την πρόσληψη νέων ε, ανθρώπων, αλλά κατανοώ το σχόλιο σας και τις επόμενες δύο εβδομάδες εμείς θα οργανώσουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τα μεγάλα διεθνή χρηματοδοτικά μέσα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με όσους έχουν προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις σε άλλες χώρες, με όσους βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι για να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες των υπηρεσίας σιδηροδρόμων, του οργανισμού σιδηροδρόμων. Έχουμε αναλάβει αυτή την προφανή δέσμευση και αυτά τα διεθνή χρηματοδοτικά μέσα νομίζω θα προσφέρουν την εμπειρία τους. Και τότε θα βάλουμε, θα στελεχώσουμε κιόλας με τα κατάλληλα άτομα. Γιατί η στρατηγική για το Δούναμπι είναι εξαιρετική για εμάς, γιατί ενισχύουμε τη συνεργασία με την Ρουμανία. και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τη βοήθεια που προσφέρουν οι Ρουμάνοι συνάδελφοι. Συνεργαζόμαστε όλο και καλύτερα. Έχουμε τα πρώτα ε, μεικτά project αυτή τη στιγμή. Η κυρία Χεσμένοβα μου έκανε την ερώτηση αυτή. Ναι, συνεργαζόμαστε με τους Ρουμάνους ομολόγους μας και αυτό ε, φαίνεται από τα δύο μεγάλα project, τις δύο γέφυρες για τις οποίες έχουμε υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης και πιστεύουμε πως εκεί θα προχωρήσουμε στα μεγάλα έργα αυτά γρήγορα. Κάτι όμως πιο αξιοσημείωτο θα ήταν αν φανταστείτε ότι στο παρελθόν μας χώριζε ο Δούναβης και ακόμα μας χωρίζει. Γιατί είναι το προφανές σύνορο μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Σε 420 χιλιόμετρα έχουμε μία γέφυρα και η Βουδαπέστη σε μία πόλη έχει 7. Όμως η νοτροπία ήταν αυτή. Αυτό μείνει στο παρελθόν και βασιζόμενοι στη στρατηγική για το Δούναβι έχουμε τα κίνητρα για να συνεργαστούμε με μεγάλα έργα τα οποία όμως να έχουν λόγο ύπαρξης και πρέπει να σου πω ότι με τους ε, Ρουμάνους μιλάμε ε, για κοινή χωροταξική ανάπτυξη των δύο όμορων περιοχών δηλαδή μέσω της γέφυρας να κάνουμε και κάποια έργα από τα Καρπάθια και να φτάσουμε μέχρι τη Βουλγαρική Θράκη με κάποια ε, project στον τουρισμό, με κάποιες άλλες αναπτυξιακές δυνατότητες. Τα κοιτάμε και θα προχωρήσουμε το συντομότερο. We have five speakers. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πέντε ομιλητές και 15 λεπτά. Παρακαλώ να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ε, χαρά μου που ήρθατε και μας είπατε τις απόψεις για την κατάσταση. Είναι αλήθεια πως τα πράγματα αλλάζουν. Ακούμε καλά νέα για μεμονωμένα προγράμματα που καιρούς καιρών, αλλά για τα θέματα τώρα απόδοσης και δυνατοτήτων υπάρχουν κάποια ερωτηματικά όσον αφορά την οργάνωση. Και το λέω αυτό ως Ευρωβουλευτής από μια χώρα που είναι καθαρός ε, ε, εισφορέας όσον αφορά τις ε, τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, για τις ε, δημόσιες δαπάνες, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες. Όταν μένει πίσω, μένουν πίσω τα προγράμματα, φυσικό είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί. Και κάποιες φορές ένα από τα προβλήματα είναι η λανθασμένη εφαρμογή των κανονισμών και των οδηγιών που σχετίζονται με τις κρατικές προμήθειες στην Ευρώπη. Ε, θα ήθελα να ακούσω λοιπόν αν προγραμματίζεται βελτιώσει όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Στόιρερ, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που προσήλθατε ενώπιον μας Ευχαριστώ και ιδιαίτερα για τον ενθουσιασμό που δείχνετε για την συνεργασία γύρω από τον Δούναβη. Ακούσαμε και λίγα λόγια για τα σχέδια της Βουλγαρίας. Πολλοί από τους συναδέλφους μου σίγουρα παρακολουθούν με ενδιαφέρον την δημοσίευση της μακροοικονομικής στρατηγικής για τον Δούναβη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την αναμένουμε με πολλές προσδοκίες και ελπίδες. Εγώ βρίσκω υποδηματικό τον τρόπο με τον οποίο η Βουλγαρία προσέγγισε το θέμα ώστε να επιταχύνει τα έργα αυτά και στο περιφερειακό επίπεδο. Με την ευκαιρία ωστόσο κύριε Υπουργέ, μία ερώτηση. Μετά από τα όσα είπε και η κυρία Κρέλ προηγουμένως. Για μένα δεν είναι άσχημο να επωφεληθεί και η ιδιωτική οικονομία από κάποια εκπαίδευση που παρέχουμε, γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε και την ιδιωτική οικονομία. Εμείς είπαμε ότι ο, οι κανόνες για τα προγράμματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αλλάξουν έτσι ώστε να μπορούν να προσλαμβάνονται και ελεύθεροι επαγγελματίες με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σας καλύπτουν λοιπόν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Το η τρίτη πτυχή της παρέμβασής μου θεωρείται ότι σε συνεργασία με περιφέρειες κατά μήκο του Δούναβη, για παράδειγμα στην Αυστρία ή στη Γερμανία, αυτό το capacity building μπορεί να γίνει γιατί και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μπορούν να διατίθεται κοινοτικοί πόροι. Αν έχετε άλλες εμπειρίες θα ήθελα να μας τις πείτε ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε, να μιλήσουμε με την Κομισιόν για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μιχαλ Πέτρου Λούχαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα που βρίσκεστε εδώ κύριε Υπουργέ σήμερα. Εγώ έχω δύο πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Το ένα αφορά την συνεργασία ανάμεσα στη Βουλγαρία και τις γειτονικές χώρες Μιλώ για τα προγράμματα διαμεθοριακής συνεργασίας με τη Ρουμανία και την Σερβία, για παράδειγμα. Πιστεύετε πως υπάρχουν αρκετά χρήματα, προβλέπονται μάλλον αρκετά χρήματα για αυτή τη συνεργασία για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί και να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής. Και δεύτερο ερώτημα αφορά επίσης τον Δούναβη. Πιστεύετε πως υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη για σημεία ενημέρωσης και εφαρμογής θεσμοί δηλαδή στις περιφέρειες, όχι μόνο συντονισμό της στρατηγικής αυτής από τις Βρυξέλλες, αλλά να υπάρχουν σημεία ε, ε συνεργασίας κατά μήκο του Δούναβη. Και αν πιστεύετε ότι αυτό είναι απαραίτητο, πώς μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Μήπως ε, καλύτερα να απαντήσετε τώρα σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για την δημιουργία δυνατοτήτων, τις και προμήθειες λοιπά. Φυσικά και έχουμε συγκεκριμένους κανονισμούς, αλλά ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Άλλο είναι να έχει κανείς όλους τους απαραίτητους κανονισμούς, νόμους τα Και, και να πούμε ότι έχουμε ενερμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και άλλο είναι το να εφαρμόζονται όλα αυτά. Να σας πω λοιπόν ειλικρινά πως η εφαρμογή εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εκμάθηση, την τυποποίηση και από τους ε, βούλγαρους δικαιούχους. Να τυποποιήσουν δηλαδή την προσέγγιση τους ε, να είναι μια ξεκάθαρη απλή προσέγγιση γιατί βλέπουμε ότι σε πολλούς τομείς υπάρχει ζήτηση, υπάρχει αυτό το αίτημα να μην γίνει μια μεγάλη δηλαδή επανάσταση στις ε, κρατικές προμήθειες, αλλά να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές ε, και ξεκάθαροι κανόνες που θα ισχύουν για όλους τους ε, δήμους και τις τοπικές αρχές. Η βουλγαρική κυβέρνηση δημιούργησε μια ομάδα εργασίας που εστίασε την προσοχή στην βουλγαρική νομοθεσία περί κρατικών προμηθειών και πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είναι καλή νομοθεσία. Ε, πρέπει όμως να τυποποιήσουμε τις διαδικασίες. Δημιουργούμε τώρα, φτιάχνουμε ε, μια νέα νομοθεσία περί κρατικών προμηθειών το 2011 το Μάρτιο. Στόχος είναι να προτείνει η κυβέρνηση τη νέα σχετική νομοθεσία αυτή ε, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα ε, τα ε, δύναμα σημεία και να βρεθούν λύσεις. Δεν θα είναι ολοκένουργος ο νόμος. Αυτός ο οποίος ήδη ισχύει είναι 100% συγχρονισμένος, δεν είναι τόσο κακός, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να, ε, ο κόσμος να το μάθει και να τυποποιηθούν οι διαδικασίες. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία, ότι σε μιλώ μαζί σας, μάλλον μακρηγορώ, αλλά γιατί καθυστερεί η Βουλγαρία τόσο πολύ με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα, σας, θα ακούσετε έλλειψη δυνατοτήτων, απορρόφησης, άλλοι θα πούνε λόγω διαφθοράς, όμως ξέρετε ποιος είναι ο πιο βασικός λόγος της αρκοπορίας μας. Είναι επειδή η Βουλγαρία το 2007 ήταν Ευρωπαίος πρωταθλητής και παγκόσμιος πρωταθλητής στις ξένες επενδύσεις κατά κεφαλή εύκολο χρήμα που πλημμύριζε τον κόσμο ήρθε στη Βουλγαρία και πολλά κτίρια, πολλά μαγαζιά ε, φτιάχτηκαν σε μια πολύ σύντομη χρονική περίοδο. Και ανάμεσα λοιπόν στο 2006 και το 2008 οι ξένες επενδύσεις ε, εισέρευσαν στην Βουλγαρία, πολλαπλασιάστηκαν κατά 4-7 ε, φορές, δηλαδή φτάσαμε στα 20 δις, ενώ ήταν συνήθως 1-2 δις οι επενδύσεις. Αυτή η διαδικασία λοιπόν μεγάλων τεράστιων προγραμμάτων, εύκολο χρήμα που πλημμύρισε τη Βουλγαρία, δεν ασχολήθηκε κανείς με τα ευρωπαϊκά ταμεία. Είναι όμως η μόνη μας σωτηρία. Γιατί αν δείτε τώρα τα νούμερα, η... από τα 9 ε, δις φτάσαμε ξανά στο 1. Ε, δηλαδή μία μείωση 10, 10 φορές μείωση και Γι' αυτό και καταλάβαμε ότι η κρίση είναι τεράστια, ότι το εύκολο χρήμα μας τελείωσε, όχι μόνο στη Βουλγαρία, όχι μόνο στην περιφέρειά μας, αλλά παντού. Και άρα πολύ υποφέρουμε από αυτό. Χρειάζεται λοιπόν η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά και κανόνες. Κανόνες, οικοδόμηση δυνατοτήτων και προγράμματα που να έχουν νόημα. Συνεχίζει στα γερμανικά η στρατηγική του Δούναβη είναι, έχει και το περιεχόμενο να διδαχτούμε από τις άλλες χώρες, όπως από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ουγγαρία και από άλλες χώρες. Να σας εκμυστηρευτώ και ένα μυστικό. Βρισκόμαστε ήδη σε επαφή με τους συναδέλφους μας ε, στην Αυστρία, καθώς επίσης στην ε, Γερμανία, στη Βαβαρία δηλαδή, κάτι το οποίο δείχνει την επιθυμία μας να είμαστε από τους πρώτους, να κάνουμε από τα πρώτα ε, κυρίαρχα έργα, τα πρώτα flagship project, Και η ασφάλεια είναι σημαντικό ε, θέμα για αυτές ε, τις χώρες και σε μια συνάντηση εργασίας με τους συναδέλφους θα συζητήσουμε για τα πρώτα έργα τα οποία θα στοχεύουν σε αυτό το θέμα κυρίως. Και γι' αυτό και η συνεργασία με τις χώρες αυτές που παίζουν ηγετικό ρόλο, που έχουν τόσα πράγματα να πούν και τόσο πολύ να μας βοηθήσουν. Έχουμε και την τεχνική αυτή βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν και πολύ ευχαριστώ ότι δεχτούμε. Έτσι λοιπόν διαμεθοριακά προγράμματα λέμε πάντοτε και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ότι τα λεφτά δεν φτάνουν ή δεν είναι αρκετά. Βλέπουμε το μακροπεριφερειακό πρόγραμμα της Αντιγικής του Δουναβή για παράδειγμα μας βοηθεί στο να αντιμετωπίσουμε ακριβώς το θέμα. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και πιστεύουμε ότι τα μακροπεριφερειακά προγράμματα ε, δίνουν και καλύτερη ευκαμψία αλλά και μια μεγαλύτερη προοπτική για να, για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε και ευρύτερους στόχους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, συνάδελφοι, ε, ξανά μάκρυνο κατάλογος, ξανά πέντε έχω. Λοιπόν, μόνο ένα λεπτό στον καθένα θα σας δώσω, λυπάμαι, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Ε, η Σοφία Κονή Λοιπόν, από ένα λεπτό ο καθένας οι επόμενοι ομιλητέ, παρακαλώ. Σαν, κελί. Σα καλωσορίζω κύριε Υπουργέ και σα ευχαριστώ για την ειλικρινή παρουσίαση και ρεαλιστική παρουσίαση σας αναφέρατε εγώ δεν θα τολμούσα να το πω αλλά είπατε ότι η βουλγαρική εικόνα έχει αμαυρωθεί και μετά περιγράψατε τις προσπάθειες που καταβάλλετε για να ε, δημιουργήσετε βιώσιμο τουρισμό και είπατε επίσης ότι θέλετε στήριξη για την ανάπτυξη περιφερειακών ε, τουριστικών ε, προϊόντων και μάρκετινγκ για τους προορισμούς σας. Πόσο δύσκολο είναι να αναπτυχθεί ο τουρισμός, ποια διαφορά υπάρχει με βάση τα χρήματα που έχετε πάρει μέχρι στιγμής για να προσελκύσετε τουρισμό ε, εσωτερικό της χώρας και εκτός της χώρας και πιο μακροπρόθεσμα ποιοι είναι οι στόχοι σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ. Προερχόμενος από το Λίντς στην Αυστρία, όντως μπορώ να πω ότι η συνεργασία με τη χώρα σας είναι ιδιαίτερα επικοδομητική και έχουμε και βιομηχάνους οι οποίοι ε, επενδύουν στη χώρα σας και έχουν πολύ μεγάλο ωφέλη και η διασύνδεση με τον Δούναβη. Θυμίζω και τη, ε, τα σκάφη Τριμαράντα, τα οποία θα ε, ε, συμβάλλουν πολύ στην επικοινωνία αυτή. Τώρα έχω ορισμένε ερωτήσεις για σας κύριε Υπουργέ. Τον Ιανουάριο διαβάσαμε ότι η Ένωση δεν ήταν ικανοποιημένη από την διαφάνεια στην καταβολή των κονδυλίων. Τι έγινε τώρα λοιπόν με τις επιστολές αυτές της Κομισιόν. Ακούσαμε ότι κάπου χάθηκαν σε κάποια συρτάρια κάποιων γραφείων και ότι δεν υπήρξε ταχεία αντίδραση από πλευρά σας. Ίσως αυτή η στάση πρέπει να αλλάξει. Αναφερθήκατε και σε μεγάλα έργα, με πολύ θετικό τρόπο, αλλά και τα μικρά έργα είναι σημαντικά και πρέπει κανείς να τα εξετάσει. αν κάποια από αυτά δεν πήγαν καλά την προηγούμενη χρονιά και χρειάστηκε να αναμένεται να παρέμβει ε, να παρέμβουν οι Βρυξέλλες ίσως μπορώ να σας θυμίσω ε, και ορισμένα θέματα τα οποία δεν μας είχαν ικανοποιήσει ιδιαίτερα. Κύριε Υπουργέ, είμαι ευτυχής που άκουσα πολλά θετικά στοιχεία, πολλές θετικές πληροφορίες, όχι μόνο για την εφαρμογή, αλλά και για τι δαπάνε, ε, τα διευθυντικά ταμεία και ε, τα κονδύλια αυτών. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να λύσετε τα προβλήματα. Είμαστε εδώ τώρα, συζητάμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά από το 2013. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για τις δικές σας προτεραιότητες στη Βουλγαρία για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Και δεύτερη ερώτηση. Έχετε προτάσεις για βελτιώσεις στο φορολογικό σύστημα. Ευχαριστώ. Ο Γευγένη Κυρίλοφ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είμαι ευτυχής που σας βλέπω σήμερα εδώ και θα πρέπει να πω ότι αξίζεται ε, κάθε δυνατή ενθάρρυνση στις προσπάθειες που καταβάλλετε για την οικοδόμηση αυτού του αυτοκινητοδρόμου που αναφέρατε. Θέλω όμως να σας δώσω μια συμβουλή. Όταν λέτε ότι το επίπεδο ήταν μηδενικό το 2007, όλοι λειτουργήσαν έτσι. Ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο του ομιλητή. Έπειτα μας είπατε για το 2008 και το 2009. Επί τη βάση λοιπόν του τι συνέβη μόνο στη Βουλγαρία δεν είναι αρκεί για να το συγκρίνουμε. Θα πρέπει να συγκρίνουμε και με τις άλλες χώρες. Και τα τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι από την 1η Οκτωβρίου. Και αυτά τα στοιχεία λένε ότι όσον αφορά τα κονδύλια της συνοχής χάσαμε. Και δεν νομίζω ότι πριν από ένα χρόνο ήμασταν τόσο χαμηλά στην απορρόφηση. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω πως ε, αξίζεται ενθάρρυνση. Ε, ε, πρέπει να φτιάξουμε διοικητικές δυνατότητες και θα πρέπει να βασιστούμε και στους βούλγαρους εμπειρογνώμονε Και με αυτά θα, τα λόγια θα κλείσω. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Το είπατε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας ότι η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική που αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό οικονομικό μοχλό για τα κράτη μας και, και, και όλος ιδιαίτερο για τη Βουλγαρία. Ξέρετε όμως και πόσο σημαντικό είναι για την Ευρώπη αυτή η πολιτική συνοχή να αξιοποιηθεί στα μάτια των πολιτών και των Ευρωπαίων συμπολιτών μας. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ποια είναι τα διαβήματα, ποια είναι τα μέσα μέσα που χρησιμοποιείται έτσι ώστε οι Βούλγαροι πολίτες να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη παρεμβαίνει, συμμετέχει στη δημιουργία υποδομών, συμμετέχει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην βουλγαρική επικράτεια ε, και πώς παίρνει αξία λοιπόν η Ευρώπη απέναντι στα μάτια των συμπολιτών σας για τα έργα που κάνει εκεί. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω και δύο λόγια στο Ρινάντο Μάλμετς που είναι επικεφαλής του τμήματος που είναι υπεύθυνο για την Βουλγαρία στην DG Regio. Ρινάλντο, παρακαλώ να είσαι σύντομος. Ε, ναι, ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Αλλά πρώτα θα πρέπει να πω ότι η επαφή με τον Υπουργό βλέπετε τον πιο αφοσιωμένο ε, υπουργό ε, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχει αναλάβει προσωπική δέσμευση ε, για, και είπε ότι αυτός ο δρόμος ήταν έτοιμος ε, εγκαίρος. Και επίσης ε, για τα Βαλκάνια λειτουργεί πολύ καλά η κατάσταση όσον αφορά τις δεσμεύσεις αλλά και τις πληρωμές. Τα κακά νέα είναι ότι μόνο 1% των κονδυλίων συνοχής στην πραγματική έχουν εκταμιευθεί και αυτό σημαίνει πως για τις μεταφορές η Βουλγαρία πρέπει κάθε μέρα να πληρώνει ένα εκατομμύριο ευρώ για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα χρήματα πριν από το τέλος της πραγματικής περίοδου. Ε, για μας ε, τα καλά νέα είναι ότι η κυβέρνηση και διάφοροι υπουργοί έχουν ε, ξεκάθαρη αξιολόγηση για την κατάσταση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και προσπαθούν να τα λύσουν. Είναι ανοιχτή η διαφάνεια, είναι κατάσταση καλύτερη και η απορροφητικότητα του συστήματος έχει αυξηθεί. Όπως σας είπα, το πρόβλημα με την πολιτική συνοχή και όσον αφορά τα μεγάλα προγράμματα και την ίσως να μην είναι αυτό τόσο πολύ σημαντικό ζήτημα για αυτή την περίοδο, αλλά σίγουρα είναι ένας μεγάλος κίνδυνος να καταλήξουμε με προβλήματα στις αρχές της επόμενης περίοδου. Δηλαδή να μην υπάρχουν αρκετά μεγάλα προγράμματα έτοιμα για την επόμενη περίοδο. Η κυβέρνηση το γνωρίζει, ο υπουργό το δουλεύει, έχει πρόγραμμα. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να αποδώσει το σύστημα. Ευχαριστώ. εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο υπουργό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού είναι πολύ σημαντικό θέμα στη Βουλγαρία. Ακόμα και φέτος, μέσα στην κρίση, η Βουλγαρία κατάφερε να αυξήσει τον αριθμό των τουριστών στη Βουλγαρία. Αυτό είναι τα καλά νέα. Το κακά νέο είναι ότι τα έσοδα ήταν χαμηλότερα. Είχαμε 2% παραπάνω τουρίστε, αλλά τα ε, έσοδα από αυτού ήταν 2% λιγότερα. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ποιου θέλουμε να στοχεύσουμε να έρθουν στη Βουλγαρία. Γιατί έχουμε την πέμπτη πλουσιότερη χώρα σε ιστορικά μνημεία. Έχουμε ένα αρχαίο κράτος στην Ένωση. Έχουμε μια χώρα που είναι σταυροδρόμι πολλών, πολλών πολιτισμών. Έχουμε ένα σωρό πράγματα να δείξουμε. Από την άλλη πλευρά όμως ε, πρέπει να δουλέψουμε για μια βιώσιμη στρατηγική Έχουμε δημιουργήσει μια ειδική επιτροπή στην Βουλγαρία. Είναι πολύ σημαντικό θέμα ο τουρισμός. Στο πρόγραμμα μας για την περιφερειακή ανάπτυξη έχουμε 150 εκατομμύρια για τον τουρισμό. Πολύ σημαντικό είναι επίσης γιατί δημιουργεί χώρο εργασίας και ποιότητα ζωής στα μικρά χωριά της Βουλγαρίας που κατά κάποιο τρόπο είχαν καταδικαστεί να ερημώσουν. Και τώρα βλέπουμε ότι η Βουλγαρία έχει 364 σπα ε, λουτρά και προσπαθούμε να φτάσουμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει στην Μαύρη Θάλασσα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά έχουμε Έχουμε 80.000 εθρακικά μνημεία, όχι μόνο στα μουσεία, αλλά έξω, στη, στη χώρα μας. Έχουμε πολύ ψηλό στόχο να αποτελέσουμε έναν προορισμό κοινό για τον πολιτισμό, το κρασί, τα λουτρά, ένα σώρο πράγματα που έχουμε στη χώρα μας και μπορούμε να προσφέρουμε. Είναι ναυσιπλοεία επίση στα γερμανικά είναι πολύ σημαντικό θέμα και το βλέπουμε και εμείς όπως οι άλλες χώρες εταίροι ε, του Δούναβη. Η ικανότητα ε, μεταφοράς μέσω του Δούναβη δεν χρησιμοποιείται παρά με, μέχρι το 8% αυτή τη στιγμή. Μέγα πρόβλημα αυτό. Εμείς συμφωνούμε μαζί σας ότι σχετικά με τη διαφάνεια μπορούμε να κάνουμε ακόμη πολλά πράγματα, αλλά σας, βεβαιώνω, σας διαβεβαιώνω για ένα πράγμα, ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα απόρριτο έγγραφο που να έχει κρυφτεί σε κάποιο σιρτάρι. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα το μέλλον της πολιτικής συνοχής και οι προτεραιότητές μας, βέβαια. Για 6 χρόνια η Βουλγαρία ήταν πραγματικά σε ένα σταυροδρόμι. Δύο από πέντε ε, αρχαίες ρωμαϊκές οδούς περνούν από τη Βουλγαρία, οι δύο Μιλιτάρικα και άλλες. Γιατί ήταν ο συντομότερος δρόμος προς την ε, Κωνσταντινούπολη, προς την Ασία, ακόμα και προς την Κίνα, ε, ταχύτατες σιδηροδρομικές διασυνδέσεις. Είχαμε μόνο μία γέφυρα, ωστόσο ε, δεν είχαμε επαρκείς αυτοκινητοδρόμους και χρειάζεται να διασυνδεθούμε με τους ε, γειτονέ μας. Για τη μεταφορά των ε, αγαθών έχουμε και πολλά αγαθά και πολλά φορτικά αυτοκίνητα και μεγάλο δυναμικό όντας στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και γι' αυτό το λόγο λέμε μεταφορές, μεταφορές και περιβάλλον γιατί η Βουλγαρία είναι ε, σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα της ενέργειας προβληματικό, προβληματική χώρα. Είμαστε ένα προβληματικό παιδί αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο και πρέπει να ε, εγγύψουμε στο θέμα αυτό της αποδοτικότητας της ενέργειας. Ελπίζουμε να, να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κονδύλια. Η Βουλγαρία σε ορισμένα όπως υπολογιστές στο business outsourcing ε, παίζει ένα σημαντικό ρόλο. εκπονούμε τώρα μια νέα στρατηγική για το εκπαιδευτικό σύστημα να ρίξει ιδιαίτερη, ιδιαίτερο βάρος σε ηλεκτρονικές τεχνολογίες και σε λεγόμενες life sciences. Μιλούμε για όλες αυτές τις προτεραιότητες, αλλά πάντως ένα πράγμα είναι σίγουρο. Αν δεν διαθέτει κανείς την βασική υποδομή ε, για τη διασύνδεσή του με άλλες χώρες, για να ε, μειώνονται οι χρόνοι ναι, δεν θα ε, υπάρχει τρόπο να αναπτυχθούμε. Βέβαια, ε, Ταμείο Συνοχή ήμασταν οι τελευταίοι, εξακολουθούμε να είμαστε στον πάτο. Δεν το κρύβουμε το γεγονό αυτό. Το Ταμείο Συνοχή είναι μέγα πρόβλημα για την Βουλγαρία. Αλλά έχουμε ένα σχέδιο και δεν θα είμαστε οι τελευταίοι ε, το 2011. Και έχουμε 7 νέα έργα στον αγωγό όπως λένε, δηλαδή θα αρχίσουν να εφαρμόζονται το 2011 και ελπίζουμε ότι δεν θα είμαστε πλέον οι τελευταίοι στην αξιολόγηση. Αλλά πάντως για την ανάπτυξη δεν είμαστε οι τελευταίοι, είμαστε μέσα στο μέσον όρο και έχουμε και πολύ φιλόδοξους στόχους. Και τέλος σας ευχαριστώ ε, Ρινάλντο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας κατανοεί, μας βοηθεί βρίσκεται στο πλευρό μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες γι' αυτό. Δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά έργα πράγματι. Έχουμε ένα πρόβλημα με ε, τον αγωγό των έργων, δηλαδή τα έργα που προωθούνται. Θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πάντως μέσα στα κακά αυτά ναι, υπάρχει και ένα καλό ότι τα τρία πιο σημαντικά έργα για τη Βουλγαρία, δηλαδή ο αυτοκινητόδρομος Χέμος, ο οποίος θα συνδέσει φτωχές περιοχές της ε, Ευρώπης, Βουλγαρία, Σερβία 1,5 δισεκατομμύριο με λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε το έργο αυτό και αυτό είναι σημαντικό, η χρηματοδότηση αυτή είναι σημαντική μέχρι το 2013. Ε, θα δείτε λοιπόν πολύ ξεκάθαρα αποτελέσματα τα επόμενα τρία χρόνια. Σας ευχαριστώ λοιπόν κυρία Πρόεδρε ε, και ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα η κυρία Χίπνερ. Σας ευχαριστούμε όλοι και όλες. Όπως είπατε, ναι, έχουμε ακόμα προβλήματα, αλλά έχουμε ένα σχέδιο. Ελπίζω κάποια στιγμή να ξαναβρεθούμε να σας ρωτήσουμε πώς πάει, ε, η εκτέλεση του σχεδίου σας. Σας ευχαριστώ για την ειλικρίνειά σας, για την ε, εικόνα που μας δώσατε και των προβλημάτων και των επιτυχιών σας και ελπίζουμε η Βουλγαρία να αποτελέσει ικανό εταίρο και για μας στην συζήτηση της μελλοντική πολιτικής συνοχής του επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ και πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε λοιπόν αμέσως στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη. Εδώ έχουμε μια δημόσια ακρόαση για την καινοτομία, της μικρομεσαίες επιχειρήσης και τη συνοχή και την πολιτική συνοχή. Παρακαλώ λοιπόν όσοι χρειάζεται να αποχωρήσουν από την αίθουσα να το κάνετε όσο δυνατόν πιο ήσυχα μπορείτε για να μην διακόψετε τη συνέχεια τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Πρέπει να σας πω πως αυτή η δημόσια κοράση γίνεται γιατί ετοιμαζόμαστε για την επόμενη περίοδο και θέλουμε καινούργιε ιδέες. Καλέσαμε για το σκοπό αυτό λοιπόν, ε, μετά από πρόταση των ομάδων, μια σειρά από εμπειρογνώμονες και θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με τον πρώτο εμπειρογνώμονα, αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ρίτζο Καινοτομία ε, και Τεχνολογικές Εξελίξεις, ο κύριος Τζον Walsh. Παρακαλώ πολύ να περιοριστείτε στον χρόνο που μας έχουμε ε, διαθέσει και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Είναι ο λόγος δικός σας. Λοιπόν, ε, Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση να ξεκινήσω εγώ τη συζήτηση. Και πρέπει να σας πω πως το να μιλάμε για καινοτομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που ήθελα να κάνω είναι για να ξεκινήσω τη συζήτηση να σας κάνω μια απογραφή του τι γίνεται στην Ευρώπη σε επίπεδο στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σήμερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτά τα στηρίζει η πολιτική για τη συνοχή. Έχω μαζί μου κάποιες διαφάνειες τις οποίες θα έπρεπε να έχετε μπροστά σας. Η στήριξη λοιπόν της επιχειρηματικότητας είναι πολύ σημαντική γιατί βοηθά πάρα πολύ είτε μέσω του προγράμματος ε, πλαίσιο για την έρευνα είτε μέσω άλλων ε, χρηματοδοτικών εργαλείων την επένδυση ε, στο χώρο των μικρομεσαίων. Και πρέπει να σου πω ότι η εξπόστη εκ των υστέρων αξιολόγηση της προηγούμενης περίοδου δείχνει πως πάνω από το 83% της στήριξης πήγε απευθείας στις μικρομεσαίες. Βλέπουμε λοιπόν και τεκμηριώνεται αυτό που στηρίζεται, ε, στηρίξαμε την δημιουργία τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου θέσεων απασχόλησης, στηρίξαμε τις επιχειρήσεις αυτές, τις οποίες επενδύσαμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε την κλασική διαφάνεια που απλώς μας υπενθυμίζει πως η πολιτική συνοχής ουσιαστικά ε, καταρχήν ε, εστιάζεται στις περιοχές σύγκλησης και αυτή η συγκέντρωση επηρεάζει το βάρος που δίδεται στη στήριξη επιχειρήσεων αλλά και στην επιλογή προτεραιοτήτων που κάνουν είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο τα κράτη-μέλη. Γιατί, χρειάζεται γιατί χρειάζεται τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν πώς θα κινητοποιήσουν αυτή τη στήριξη. Στην επόμενη διαφάνεια έχω απλώς κάποια στοιχεία. Αφήστε στην άκρη τα μεγάλα ποσά και για την καινοτομία να δείτε. 25% της πολιτικής συνοχής επενδύεται στην ε, καινοτομία, στην ευρύτερη καινοτομία. Είναι λοιπόν 86, το 25% των 86 δισεκατομμυρίων. Το 45, λοιπόν, 45 δις πηγαίνει στην καινοτομία και 55 δις πηγαίνουν στις επιχειρήσεις. Ένα 16% λοιπόν. Και λέμε πως 40, 45 δις, επαναλαμβάνω, τη στήριξη επιχειρήσεων ε, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως στήριξη στην καινοτομία. Δηλαδή το 25% όπως σας είπα του συνολικού προϋπολογισμού. Στα 55 δις για τις επιχειρήσεις ξέρουμε πως τα 27 από 7, δηλαδή το ίμιση, διατίθεται αποκλειστικά και μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βλέπετε το τυράκι στη διαφάνεια και ένα μεγάλο τμήμα πηγαίνει στον κλάδο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, κυρίως στις οικολογικές ε, καινοτομίες, στην καλύτερη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής, όπως επίσης και στην εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, τα γνωστά startup, εκεί το χρηματοδοτικό μέσο μας έχει μεγάλο ε, μεγάλη δράση, ε, κυρίως μέσω κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου. Μην προσθέσετε αυτά τα 86, 55 και 27 δις, γιατί μιλάμε για υποκατηγορίες. Με μία εξαίρεση υπάρχουν κάποιες κατηγορίες στήριξη επιχειρήσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον ε, τίτλο ή υπό τον τίτλο της καινοτομίας. Αυτές οι κατηγορίες συνδέονται με μη κλαδική χρηματοδότηση, με δανειοδότηση και με επένδυση σε ε, υποδομές επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τμήμα του προεκπλογισμού που δεν ε, πηγαίνει στην καινοτομία. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε πως έχουμε κάποια σχόλια για τις στάσεις της επενδύσεις στην καινοτομία. Σας μίλησα λοιπόν για 25% προηγουμένως πρόκειται να τελειώσουμε, να κλείσουμε σύντομα μία συνοπτική ανακεφαλωτική έκθεση για τις δράσεις μας στην καινοτομία και εκεί διαπιστώσαμε πως υπήρξαν τρεις άξονες, τρεις βασικοί άξονες στήριξης καινοτομίας. Πρώτα απ' όλα, περιβάλλονται φιλικά προς την καινοτομία και το χρήστη. Θα σας δώσω για τις μικρομεσαίες αργότερα κάποια παραδείγματα Δεύτερον, τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες στηρίζουν την εφαρμοσμένη ε, έρευνα, τμήμα της δικής μας πολιτικής συνοχής, όχι μόνο λοιπόν ε, θεωρητική αλλά και εφαρμοσμένη έρευνα και κυρίως εφαρμοσμένη και τρίτον μεταφορά γνώσης και δημιουργία ε, κόμβων καινοτομία τα γνωστά clusters. Πολύ σημαντικά αυτά, τα βρίσκεται σε διάφορα κράτη-μέλη. Βλέπετε όμως να κυριαρχούν και συγκεκριμένα είδη στήριξη, είτε σε περιοχές ανταγωνιστικότητας, είτε σε περιοχές σύγκλησης. Αυτό λοιπόν ενισχύει την άποψη το ότι ο τρόπος με τον οποίο τα μέτρα καινοτομία και στήριξης των επιχειρήσεων κινητοποιούνται διαφέρουν αρκετά από χώρα σε χώρα. Μία τάση που διαφαίνεται είναι οι τελευταίες δύο τελίτσες. Κοιτάξτε το έγγραφο γιατί εγώ δεν βλέπω να σας το διαβάσω. Είναι πως έχουμε δύο γενικές τάσεις. Καταρχήν εστιάζουμε, συγκεντρώνουμε αυτά τα κονδύλια στους κόμβους αυτούς, στα κέντρα αριξίας, ε, στην τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη και το δεύτερο είναι πως θέλουμε να εμπλέξουμε περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην καινοτομία, να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες στήριξης και πλαισίωσης αυτών μέσω των κόμβων, των κλάστερ που μας διευκολύνουν να μετακινηθούμε προς μια κοινωνία της γνώσης με την ευρύτερη έννοια. Άρα λοιπόν οι διαδικασίες, ο σχεδιασμός και όχι μόνο η καθαρή καινοτομία μας ενδιαφέρουν. Στην επόμενη διαφάνεια σας δίνω κάποια παραδείγματα. Και θα έλεγα όχι ακριβώς παραδείγματα, αλλά εδώ είναι οι έξι κατηγορίες στήριξη μικρομεσαίων. Οι δύο πρώτες στην μελέτη την οποία πρόκειται όσον ούπο να δημοσιεύσουμε σχετίζονται με τα περιβάλλοντα τα οποία είναι φιλικά προς τις επιχειρήσεις, δηλαδή υπηρεσίες πληροφορικής, πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφορικής από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μετά Έχουμε και τρεις κατηγορίες που απευθύνονται περισσότερο και συνδέονται περισσότερο με την βελτίωση των τεχνικής εκμετάλλευσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή η οικολογική καινοτομία για παράδειγμα, ε, πρόσβαση στην έρευνα για τις μικρομεσαίες και τρίτον η κοινωνία της γνώσης εκεί Πολλά κονδύλια στην Ευρώπη έχουν επενδυθεί μέσω του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα, μέσω των δικτύων των επιχειρηματικών, μέσω των κλάστερ και μέσα βεβαίως, μέσω βεβαίως του κοινωνικού ταμείου για τις ε, καινούργιες επιχειρήσεις, τις startup. Στην επόμενη διαφάνεια, μία από τις τελευταίες που θα σας δείξω, ήθελα να σας δείξω τις διαφορές ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη η στήριξη και η κινητοποίηση των διαφορετικών ταμείων γίνεται με διαφορετική ένταση στα διάφορα κράτη και μιλάμε κυρίως για το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και για το κοινωνικό ταμείο. Κοιτάξτε, δεξιά έχουμε τις τρεις τελευταίες στήλε. Βλέπετε πως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των 15, ε, όπου η στήριξη έχει φτάσει στο 11%, ε, με συγχωρείτε, η στήριξη των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το 11% της ε, συνολικής χρηματοδότησης, ενώ δίπλα που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών, εκεί, με συγχωρείτε, στις, Ευρωπαϊ... στις καινούργιες χώρες, στα 12 κράτη, είναι μόλις το 5%. Τι συμβαίνει λοιπόν στα νέα κράτη τα οποία είναι όλα σχεδόν περιοχές σύγκλησης. Έχουμε πολλά κονδύλια που πάνε στις υποδομές, και τα ποσά που κρύβονται πίσω από το 5% της επιχειρηματικής στήριξης είναι μεγάλα. Τουλάχιστον σε σχέση με παλαιότερες δράσεις αντίστοιχες σε αυτά τα κράτη. Αλλά ακόμα και στα πιο παλιά κράτη-μέλη βλέπετε υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση της έντασης ή του ρυθμού με τον οποίο στηρίζονται οι επιχειρήσεις. Και βέβαια εξαρτάται και από τις έξι κατηγορίες τις οποίες παρουσιάσα στην προηγούμενη διαφάνεια και το πώς αυτές συνδυάζονται μεταξύ τους. Τώρα, η έκθεση στρατηγικής, αν θέλετε περισσότερες προφορίες για, την, για τον ρυθμό προόδου αυτών των μέτρων, να σας πω πως η στήριξη επιχειρήσεων γενικά έδειξε μία επιλογή, ένα αριθμό επιλογή τη τάξη του 23% για τα τέλη του 2009, φαίνεται από την έκθεση του Μαρτίου τη Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαφέρει ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτέ τι προφορίε μπορείτε να τι βρείτε στην ιστοσελίδα μα, μάλλον στον ιστοτοπό μα. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι πω τα υπόλοιπη κωδική στήριξη επιχειρήσεων που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το μέγεθος των επιχειρήσεων, τα υπόλοιπα 28 δις, έχουν μεγαλύτερη ε, με γρηγορότερο ρυθμό ανάληψης υποχρεώσεων. Δηλαδή είναι στο 37% και όχι στο 23%. Νομίζουμε πως αυτό εξηγείται από το εξή. Ε, τα καινοτόμα μέτρα με πολύ αργό τρόπο και κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα χρησιμοποιούν οι μικρομεσαίες. Και μάλιστα ίσως χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους χρηματοπιστωτικής στήριξης μέσω των μη κλαδικών ή των μη, ε, μη κλαδικών ε, εργαλείων χρηματοδότησης ή μέσω των μέσων που δεν ε, καθορίζονται ή που δεν απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένα μεγέθη. Έχουμε λοιπόν τα μη κλαδικά ή τα λιγότερο κλαδικά, τα οποία προσφέρονται, είναι ανοιχτά σε όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Και με συγχωρείτε που διαφημιζόμαστε τώρα, αλλά έχουμε εμείς τους τελευταίους, το τελευταίο διάστημα παρουσιάσει αυτές τις θερμοκοιτίδες καινοτομία ή αντιδραστήρες καινοτομία, όπου κάνουμε κάποι, δίνουμε κάποιες πληροφορίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν. Μπορώ να σας δώσω τις πληροφορίες αργότερα και έχουμε και μία σειρά μέτρων στο δεύτερο link λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια θα δείτε παραπάνω από 50 παραδείγματα στήριξης επιχειρήσεων για διάφορα είδη καινοτομίας από όλη την γάμα δραστηριοτήτων που στηρίζουν τις επιχειρήσεις. Ελπίζω να τα βρείτε χρήσιμα. Και να είναι μια καλή εισαγωγή ε, αναμένω λοιπόν τις υπόλοιπες παρουσιάσεις και την συζήτηση που θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στον κύριο Μπερντελόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα να ρίξω ιδιαίτερο ε, φως σε ένα τμήμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δεν είναι πάντα το, τόσο γνωστέ στο κοινοτικό επίπεδο, δηλαδή οι μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει ε, στο βιοτεχνικό τομέα, που καμιά φορά είναι ιδιαίτερα και Στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε, υπενθυμίζω μάλλον, ότι επί 21 εκατομμυρίων 98,5% ε, είναι, πολύ, είναι μικρές επιχειρήσεις και 92% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικροεπιχειρήσεις. Ο, η διαδικασία της καινοτομίας σε αυτές τις μικρές και μικροεπιχειρήσεις είναι μια διαρκής διαδικασία από μια καινοτομία που είναι ε, σύμφωνα με την ε, ζήτηση είτε των προμηθευτών είτε των καταναλωτών. Αυτή την καινοτομία τη βρίσκει κανείς και στη χαμηλή τεχνολογία και στην υψηλή τεχνολογία σύμφωνα με τις ανάγκες των αγορών, σύμφωνα με, ε, με την κατανομή έργου αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν πολλές μικρές και μικροεπιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν και στον τομέα της ε, υψηλής τεχνολογίας. Άκουσα συχνά ότι οι μικροεπιχειρήσεις δεν είναι ικανές να ε, κάνουν έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Ωστόσο, τις βρίσκουμε στην νανοτεχνολογία, στις επικοινωνίες, ακόμα και στην τεχνολογία του διαστήματος και του πλάσματος όπου βρίσκει κανείς πολλές μικροεπιχειρήσεις με λιγότερο από 10 ε, εργαζομένους και στον εξωτερικό τομέα που ε, καινοτομούν στον τομέα της ενέργειας και την συμπαραγωγή ενέργειας. Δύο χαρακτηριστικά. Είναι σημαντική διασπορή, δηλαδή προ, προωθούν και περαιτέρω τις ε, ενέργειες αυτές και τους επιτρέπει να περάσουν τις νέες καινοτομίες τελικά στους καταναλωτές με μια φάση καινοτομία που προσαρμόζει τι καινοτομίες αυτές στην αγορά και στη ζήτηση. Άλλο σημαντικό είναι ότι οι ίδιες αυτές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ξεκινούν δηλαδή καινοτόμε καινοτόμες σε όλους τους τομείς ε, της οικονομικής δραστηριότητας, ακόμα και της πολύ υψηλής ε, τεχνολογίας. Κάτι άλλο που πρέπει να τονίσω είναι η σημασία της πράσινης οικονομίας ό,τι έχει σχέση με την κατασκευή, με την οικοδομή, με την διαχείριση της ενέργειας σε όλες τις ευρωπαϊκές σχεδόν περιφέρειες βρίσκει κανείς καινοτομίες που προέρχονται από τις μικρές ή τις μικροεπιχειρήσεις. Τρίτο, οι συνέπειες που έχουν οι ενέργειες των επιχειρήσεων αυτών και για την κοινωνική συνοχή επιτόπου, εδώ τονίζω δύο πράγματα οι μικρές και μικροεπιχειρήσεις που καινοτομούν δεν συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα ή τους μεγάλους πόλους. Τις βρίσκει κανείς παντού, ακόμα και στην Ήπεθρο, ακόμα και στις μειονεκτικές περιοχές, όπου υπάρχουν πολλές μικροεπιχειρήσεις, πολύ καινοτόμε και στην υψηλή τεχνολογία που βρίσκονται ακόμα σε ορεινές περιοχές, στις νησιωτικές περιοχές και που πολύ συχνά οι επιχειρήσεις αυτές θα έλεγα ότι η καινοτομία δημιουργεί απασχόληση και μάλιστα απασχόληση και επιτόπου που, έχουν και, που έχει και χαρακτήρα σταθερότητας. Τρίτο χαρακτηριστικό είναι η χρηματοδότηση. Εδώ υπάρχει ένας μικρός πίνακας κατανομής των χρηματοδοτήσεων ανά μικρές επιχειρήσεις. Κυρίως είναι ήδη πόροι και ε, ενισχύσεις δημόσιες ή περιφερειακές σχετικά απούσες είναι οι τράπεζες και αρκετά απόν είναι και το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Άρα έχουν κάποιες δυσκολίες πρόσβαση στα ταμεία αυτά οι επιχειρήσεις αυτές, όπου αναπληρούνται όμως από τις περιφερειακές ενισχύσεις και με τον τρόπο αυτό και το Περιφερειακό Ταμείο ενισχύει. Σημαντική επίσης είναι η παροχή ε, συμβουλών από τις ενδιάμεσες τις διαμεσολαβητικές οργανώσεις, διότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην καινοτομία αν δεν έχουν την συνοδεία των διαμεσολαβητικών αυτών οργανώσεων. Τα προβλήματα τώρα είναι πέντε βασικά. Πρώτο, δεν υπάρχει καμία οικονομική ανάλυση ή στατιστική στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο ε, επίπεδο των χωρών μελών σε ό,τι αφορά την σημασία στην καινοτομία των μικρών και μικροεπιχειρήσεων. Δεν ξέρουμε αυτό το 90 των επιχειρήσεων τι ε, συνέπειες έχει η δραστηριότητά του. Έχει δοθεί εξάλλου σημαντική ε, προτεραιότητα στις υψηλές τεχνολογίες, τεχνολογίες εχμής, στις ε, τεχνολογίες με ταχύτατη ανάπτυξη, αλλά λησμονούνται συχνά όλες οι καινοτομίες που θα έλεγα τρέχουσες. Μία από τις μεγάλες προτεραιότητες που δίνονται στις καινοτόμες επιχειρήσεις και τον Δεκέμβριο του 2008 το ε, Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνισμού είχε ζητήσει να ανοιχθεί η πολιτική ανταγωνισμού για τις ε, μικρές και μεσές επιχειρήσεις τις καινοτόμες. Ε, τρίτος παράγοντας είναι αυτό που λένε στα αγγλικά sleeping innovators. Αυτοί, αυτές δηλαδή οι καινοτόμες επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται, που υπάρχει ένα περίπου 5% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι τέτοιοι sleeping innovators. Έχουν δηλαδή ικανότητα, έχουν καινοτόμα ικανότητα, αλλά δεν ξέρουν καν ότι εφευρίσκουν νέα πράγματα. Ένα περίπου εκατομμύριο, εκατομμύριο επιχειρήσεων που είτε λόγω έλλειψης παρακολούθησης είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης δεν κάνουν καν το βήμα να προχωρήσουν σε συνεργασία ε, με άλλες οργανώσεις ώστε να δώσουν ε, σάρκα και οστά σε κάποιες καινοτομίες. Και τέλος ε, το πρόβλημα της κουλτούρας, της νοοτροπίας δηλαδή της επιχείρησης και της καινοτομίας που συχνά το δημόσιο δεν έχει αρκετή ιδέα του ρόλου, του καινοτόμου ρόλου που μπορούν να παίξουν αυτές οι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και δεν μιλώ βέβαια καν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δίνουν κυρίως τον καινοτόμο χαρακτήρα στις μεγάλες ή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους και ε, παραγνωρίζουν, δεν προβάλλουν καθόλου δηλαδή, το καινοτόμο έργο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που είδαμε στι αναλύσει μα είναι ότι οι επιχειρήσει αυτέ έχουν σημαντικό πρόβλημα πρόσβαση στην πιστοποίηση, η οποία έχει γίνει συχνά ένα φραγμό για την πρόσβασή του στις αγορέ, διότι είναι πολύ δύσκολο για τι επιχειρήσει αυτέ ε, να ε, καταθέσουν αιτήσει ευρεσιτεχνία και να επιτύχουν την διαπίστευση του προϊόντος τους. Ο ρόλος τώρα της πολιτικής της συνοχής, ποιος είναι. Αυτά που γνωρίζουμε από τις μελέτες που έχουμε κάνει στον χώρο των μικρών και μεσών επιχειρήσεων είναι ότι ο ρόλος της περιφέρειας είναι πολύ σημαντικός. Ένα, περίπου το 90% των ε, ευρωπαϊκών περιφερειών παρεμβαίνουν για να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Κατά μέσον όρο, 7 κατηγορίες παρεμβάσεων, πρώτα με πόλους καινοτομίας και κέντρα διασποράς, Δεύτερο, θα επανέλθω αν θέλετε σε αυτό, προγράμματα παρακολούθησης και παροχή συμβουλών για την καινοτομία. Τρία κυρίως μέτρα στην ανακάλυψη κυρίως αυτών των sleeping innovators και της καινοτόμου ικανότητας των επιχειρήσεων. Άλλο σημαντικό είναι η βοήθεια για να επιτύχουν την ε, ε, πιστοποίηση των προϊόντων τους με διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ. Και αυτό σημαντικό. Τα άλλα σημαντικά θέματα είναι, δηλαδή της παρέμβασης των περιφερειών, είναι συχνά η υποστήριξη των εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και κέντρων ε, διασποράς της καινοτομίας, επίσης η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά, η εκπαίδευση και επίσης ειδικέ χρηματοδοτήσεις από τις ίδιες τις περιφέρειες με την δημιουργία ε, ειδικών κεφαλαίων ανάληψης κινδύνου που να δίνουν τραπεζικές εγγυήσεις ειδικά για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι συνήθως τα ίδια, ότι δεν έχει γίνει καταστεί ακόμα δυνατόν στο επίπεδο των ε, ε, χωρών μελών να εντοπιστούν οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είναι καινοτόμες. Οι περιφέρειες το γνωρίζουν αλλά δεν έχει γίνει ειδικά δουλειά γι' αυτό και ιδίω οι ευρωπαϊκοί δείκτε σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Οι τρει δείκτε που αναφέρονται στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσεις, όλοι αυτοί οι δείκτε αναφέρονται στι επιχειρήσει τη άνω των 10 εργαζομένων. Τι γίνεται με αυτέ που είναι κάτω από του 10 εργαζομένου. Δεύτερο πρόβλημα, όταν εξετάζει κανεί του δείκτε ε, των ανθρώπινων πόρων και οι τρει αυτοί ε, δείκτε αναφέρονται σε πανεπιστημιακά πτυχία δεν μιλούν καθόλου για ικανότητες ή γνώσεις επαγγελματικές που βοηθούν ωστόσο στην ανάπτυξη αυτής της καινοτομίας. Πολλοί από τους επαγγελματίες, πολλοί από τους επιχειρηματίες έχουν επίπεδο προσόντων πάρα πολύ υψηλό που τους επιτρέπει οι ίδιοι να είναι καινοτόμοι. Πάλι ε, δεν υπάρχει απολύτως καμία αναφορά στο κοινοτικό, στο ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή, των ικανοτήτων αυτών, των επαγγελματικών ικανοτήτων κάτω από το, Ευρωπα... από το ε, Πανεπιστημιακό Πτυχίο. Δεν υπάρχει καμία ανάλυση επίσης ότι αφορά τις επιπτώσεις των διαθροτικών ταμείων. Στις αναλύσεις που έχουμε κάνει και διαβιβάσει διαπιστώνουμε ότι το πολύ 1, 2 ή 3% των μικρών επιχειρήσεων εποφελούνται από τα διορθωτικά ταμεία. Το ίδιο για τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι η σύγχυση μεταξύ των ε, κοινοτικών κονδυλίων. Δεν υφίσταται συνέργεια μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα διαθωτικά ταμεία, περιφερειακά, ε, διάφοροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Μία μικρή επιχείρηση μόνη της χάνεται, ε, τελεί εν συγχύση ανάμεσα σε όλες αυτές τις δυνατότητες. Όταν λοιπόν υπάρχει μια πρωτοβουλία σε θέμα καινοτομίας θα πάει στον πρώτο της χανεται τελει εν συγχυση αναμεσα σε ολες αυτες τις δυνατοτητες οταν λοιπον υπαρχει μια πρωτοβουλια σε θεμα καινοτομία, θα παει στον πρωτο τη συνομιλητη που είναι η περιφέρεια. Τέλος, οι πραγματικότητες της διοίκησης. Δηλαδή πάλι εκεί υπάρχει ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων των επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων και αυτών που λαμβάνουν τις πολιτικές εν τέλει αποφάσεις. Τελευταία διαφάνεια. Με ρωτήσατε λοιπόν ποιες είναι οι δυνατότητες για μετά το 2013 νομίζω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτεί κανείς κάθε ε, ίχνος ε, καινοτόμου δυναμικού που υπάρχει στην κοινότητα. Αυτό που κάνει οι Αμερικανοί με το πρόγραμμα σπάε, Βοήθεια, παροχή συμβουλών και ανάπτυξη, πρόθεση στην αγορά. Η κοινοτική πολιτική δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του υφιστάμενου δυναμικού, γιατί κυρίως στοχεύει στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχει λοιπόν ε, το Small Business Act, το οποίο επιτρέπει ωστόσο την ανάπτυξη αυτή. Τώρα, προτείνονται ορισμένες προτεραιότητες. Πρώτα, μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική της καινοτομίας για τις μικρές και για τις μικροεπιχειρήσεις. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να φροντίσουμε ώστε αυτή η smart specialization που γίνεται και μέσω της επικοινωνίας της ευρωπαϊκής πολιτικής για την καινοτομία να μην αποκλείει άλλες επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται σε αυτόν τον ειδικευμένο τομέα. Δεύτερη προτεραιότητα επίσης πολύ σημαντική οι ενδιάμεσες οργανώσεις. Αν δεν συνεργαστούμε με τις ενδιάμεσες οργανώσεις αποκοβόμαστε από όλο αυτό το φάσμα των ε, καινοτόμων επιχειρήσεων. Άλλο είναι να ευνοήσουμε την το συνδυασμό των προσπαθειών μεταξύ των επιχειρήσεων και αυτών που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Επίσης, προσαρμογή και συντονισμός των ε, οικονομικών μηχανισμών, των χρηματοδοτικών δηλαδή ε, μηχανισμών. Να υπάρξει μια διευκρίνηση, ένα ξεκαθάρισμα των μηχανισμών αυτών που να διευκολύνει την παροχή υποστήριξης ε, προς τις επιχειρήσεις αυτές. Πέμπτη προτεραιότητα, θα ήθελαμε να προτείνουμε δηλαδή μια ευρωπαϊκή εκστρατεία για την ανακάλυψη αυτών των λεγόμενων sleeping innovators, των μικρών αυτών καινοτόμων επιχειρήσεων που υπνώτουν κατά κάποιο τρόπο. Επίσης θέλουμε μια εργασία ενημέρωσης, διότι δυστυχώς οι περιφέρειες μόνες τους δεν γνωρίζουν η αριστερά τους τι πει η δεξιά τους σχετικά με τις επιχειρήσεις αυτές. Εγώ ήρθα σε επαφή με πολλές περιφέρειες και μου είπαν ότι σε ακτίνα 200 χιλιόμετρων δεν γνωρίζουν τι κάνουν οι διάφορε επιχειρήσει. Άλλο είναι ε, να δοθεί εκπαίδευση στο προσωπικό για αυτήν την οτροπία τη καινοτομία. Ε, να διευκολυνθεί επίση, ε, last but not least, όλε οι πολιτικέ που μπορούν να θεσπιστούν δεν θα έχουν πολλά αποτελέσματα εάν δεν υπάρξει μια πραγματική απλούστευση των διαδικασιών για την πρόσβαση σε κοινοτική χρηματοδότηση. Όλοι όλοι βεβαίως μιλούν γι' αυτό. Έχουμε δώσει ένα έγγραφο πολλών προτάσεων και των ενδιαφερομένων και των επιχειρήσεων για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων και των καινοτόμων ιδίως επιχειρήσεων στις χρηματοδοτήσεις αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας και για τις ιδέες σας και τώρα θα θα περάσουμε στον κύριο Μάισινς από το Δυτικό Μπραμπάντ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι διευθυντής της, ε, του Οργανισμού Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, του Δυτικού Μπραμπάντ. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ε, η ε, το Διοικητικό μας Συμβούλιο είναι οι τοπικές αρχές και τα μέλη της επιχειρηματικής μας κοινότητας. Και έχουμε δύο πολύ σημαντικά ε, βασικά καθήκοντα. Να συμβάλλουμε στην ε, το περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Αυτό το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Καταρχήν να συμβάλλουμε στηρίζοντας τις επιχειρήσεις για για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης προσπαθούμε να προσελκύσουμε νέους επενδυτές στην περιφερειά μας και το τρίτο μας καθήκον είναι η σύνδεση με αυτήν όλη την ομάδα. Προσπαθούμε μέσω προγραμμάτων να ενισχύσουμε την οικονομική δομή της περιφέρειας. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Σε αυτό το, τη διαφάνεια βλέπουμε πως ο κόσμος είναι σε μεταβατική περίοδο και στην δική μας περιφέρεια πρέπει να αντιμετωπίσουμε την οικονομική μετάβαση. Έχουμε μια προσέγγιση λοιπόν οικονομική και σε σχέση, σε σύνδεση με το οικοσύστημα της περιοχής. Πού βρισκόμαστε εμείς και ποια είναι η σχέση μας με τις κάτω χώρες. Είμαστε ανάμεσα στα δύο μεγάλα λιμάνια, το Ρότερνταμ και την Αμβέρσα. Και αυτό έχει δώσει στην οικονομική μας ανάπτυξη την κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα. Η μετάβαση που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι η παραδοσιακή βιομηχανία και η γεωργική βιομηχανία ε, βρίσκεται σε μια ύφεση. Και ε, τώρα έχουμε την ε, αύξηση των γραφείων και των ευρωπαϊκών κέντρων διανομής, κυρίως μέσω της Αμβέρσας και του Ρότερταμ, των μεγάλων αυτών ευρωπαϊκών λιμανιών. Δεν έχουμε μεγάλα κεντρικά γραφεία και δεν έχουμε τεχνικό πανεπιστήμιο. Μπορούμε να δούμε δηλαδή την περιφέρειά μας ως μια μέση περιφέρεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμάστε. Διότι στην περιφέρειά μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε ακολουθήσει μια ειδική προσέγγιση. Επιλέξαμε για την περιφερειακή αντιπρόσωπη, ε, ανάπτυξη συγγνώμη, να έχουμε τρεις βασικούς άξονες, τρεις πολύ σημαντικούς τομείς, στον τομέα της συντήρησης, που δουλεύει για τη μεταπαιδευτική βιομηχανία, έπειτα οικονομία βασισμένη στα βιολογικά προϊόντα, είναι μια οικονομία η οποία έχει τεράστια ανάπτυξη στην περιοχή μα και έπειτα έχουμε και την τεχνική υποστήριξη, logistics. Αυτοί είναι οι τρει τομείς στου οποίους εστιάζουμε την προσοχή μας. Στις κάτω χώρες έχουμε μια νέα πολιτική που εγκαινιάστηκε το 2010 και λέμε, την ονομάζουμε ε, πολιτική των ε, εχμών στη Δέλτα, δηλαδή των ε, πιο βασικών μας ε, οικονομικών τομέων. Και έχουμε βάλει Γι' αυτό χρήματα όχι μόνο η εθνική κυβέρνηση αλλά και οι ε, τοπικές ε, αρχές. Πολλά χρήματα δηλαδή ε, σε συνδυασμό με τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής. Ποια είναι τα αποτελέσματα της τετραετούς αυτής πολιτικής που έβαλε 592 εκατομμύρια ευρώ στην πολιτική αυτή. Ποια είναι τα αποτελέσματα. Ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι οι επιχειρήσεις αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα κέρδισαν 1,2 δις ευρώ χάρη σε αυτή την πολιτική. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα σε εθνική κλίμακα. Εδώ έχουμε μια αξιολόγηση της πολιτικής μας για ε, το εθνικό επίπεδο. Βλέπετε ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Η νέα αυτή προσέγγιση δηλαδή λειτουργήσε πολύ καλά. Ε, είχε ως αποτέλεσμα πολλές νέες υπηρεσίες και απόδοση, καθώς και μια όθεση σε καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο. Και θα ήθελα να σας δείξω τα αποτελέσματα για το νοτιοδυτικό κομμάτι. Έχουμε λοιπόν αποτελέσματα ήδη για τέσσερις ε, βασικούς τομείς. Ο ένας είναι η τεχνική υποστήριξη. Καταφέραμε να έχουμε αυτό τα αποτελέσματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έφτασε στην περιφέρειά μας ένα Ολλανδικό Ινστιτούτο για προηγμένη τεχνική υποστήριξη και μπόρεσε να επιταχύνει την καινοτομία στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης καθώς και ειδικά ε, ειδικού ε, εκπαιδευτικούς πυλώνες που έχουν σχέση με τον τομέα. 7 προγράμματα συνεργασίας με 49 επιχειρήσεις του τομέα της τεχνικής υποστήριξης και οι περισσότερες από αυτές είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν στόχο την καινοτομία. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Τώρα, ο δεύτερος σημαντικός τομέας είναι η συντήρηση. Συντήρηση όπου υπάρχει χωριστός εκπαιδευτικός κλάδος για τη συντήρηση στην από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι και το πανεπιστήμιο. Ένας νέος επαγγελματικός τομέας και σχετικές σπουδέ θεσπίστηκαν μέσα σε τέσσερα χρόνια. 11 προγράμματα διοργανώσαμε για την ε, βιομηχανία της συντήρησης με 223 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και επίσης ο κλάδος αυτός αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα δικό του βραβείο ε, και σήμα το αποκάλεσε συντήρηση παγκόσμιας κλάσης για να δείξει τη σημασία και την αριστεία του τομέα στη χώρα μας. Έχουμε ε, τώρα για τον άλλο τομέα της οικονομίας που βασίζεται στα βιολογικά προϊόντα, έχουμε επίσης 7 ε, προγράμματα συνεργασίας. Τώρα, οι στόχοι μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια καταφέραμε η περιφέρειά μας να μπορεί να κάνει τη δική της στρατηγική ατζέντα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Και αυτό που θέλουμε είναι να προχωρήσουμε περισσότερο στους σε άλλους ε, σε αυτούς τους τρεις τομείς, ώστε να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Να μην ε, παρακμάσουν δηλαδή λόγω της παγκόσμιας ε, οικονομικής κρίσης. Στόχος είναι ότι οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι να παραμείνουν στην περιοχή μας. Επόμενη διαφάνεια, αυτό που θέλουμε επίσης να πετύχουμε ε, στην περιφερειακή κλίμακα, στην περιφέρειά μας, είναι να έχουμε τις απαραίτητες υποδομές για αυτούς τους τρεις τομείς. Δηλαδή, ε, Ινστιτούτα Εχμής, ε, πανεπιστήμια, ερευνητικές εταιρείες και θέλουμε να, έτσι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως φυτόρια για, αυτόν τον, για αυτούς τους τρεις τομείς. και επίσης να δημιουργήσουμε τρεις νέους εκπαιδευτικούς πυλώνες, έναν για κάθε έναν από τους τρεις κεντρικούς μας τομείς. Και αυτό σημαίνει νέες επενδύσεις στους τρεις αυτούς τομείς. Να οθήσουμε δηλαδή την ε, πολιτική μας μέσω αυτών των τριών βασικών ε, κλάδων. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια είναι να έχουμε ένα κάμπους ε, για την αλυσίδα παροχή στην Πρέντα, ένα, ε, το Ολλανδικό Ινστιτούτο για την Συντήρηση Παγκόσμιας Κλάσης στην Πρέντα, ε, ένα ειδικό πανεπιστήμιο για την συντήρηση αεροσκαφών, καθώς και ένα κέντρο πυροχνομοσύνης για την οικονομία που βασίζεται στα βιολογικά προϊόντα. Ε, θέλουμε να ρεστεύσει επίσης το, το τμήμα της ε, πράσινης χημία που ήδη είναι βασισμένο, ιδρεύει μάλλον στο Bergen Zom, καθώς και να ελκύσουμε επενδυτέ στην περιφέρειά μας. Τέλος, αυτό που θέλω να τονίσω σήμερα εδώ είναι ότι είναι δυνατόν σε μία μέση περιφέρεια να βελτιωθεί ε, και να προωθηθεί η καινοτομία των μικρομεσαίων μέσω της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, με τους εκπαιδευτικούς κύκλους και την κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Ε, δίνει μια επιπλέον ισχύ και συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας ε, παγκοσμίω. Μια τελευταία διαφάνεια όπου ε, έχουμε, αναφέρω κάποιους προβληματισμούς που θα μπορούσαμε να τους σκεφτούμε, θα μπορούσαμε να μας απασχολήσουν. Ε, όταν επιλέγουμε μια τέτοια προσέγγιση με βασικούς κεντρικούς τομείς, κεντρικούς άξονες, θα πρέπει να μετακινηθούμε από τη στήριξη σε μεμονωμένα προγράμματα στην στήριξη στρατηγικών περιφερειακών προγραμμάτων. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος εργασίας. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι όταν αυτό προσαρμόζεται στην ε, περιφερειακή προσέγγιση λοιπόν, θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων ετών χρειάζεται ισχυρή κυβερνητική ε, στήριξη. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να ε, ξεκινήσει όλη αυτή η προσπάθεια. Επίσης, για να μπορέσει κανείς να συνεργαστεί με τις επιχειρήσεις και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χρειάζονται χρήματα για να λειτουργήσει η συνεργασία. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, ε, από την εμπειρία μου, είδα ότι οι θύνοντες για τη λήψη των αποφάσεων δεν το αναγνωρίζουν αυτό το στοιχείο. Δηλαδή πιστεύουν ότι η συνεργασία από μόνη της θα γίνει. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Πρέπει δηλαδή να καταβληθεί η προσπάθεια και να δαπανωθεί χρήμα για να έχει κάνει τα αποτελέσματα που σας έδειξα. Τελευταία παρατήρηση που θέλω να αναφέρω είναι η διατομιακή προσέγγιση. Έχουμε παρατηρήσει στην περιφέρειά μας ότι οι επιχειρήσεις ε, δημιουργούν δίκτυα βασικά στο δικό τους κλάδο και στη δική τους αλυσίδα. Όταν όμως ε, μιλάμε για ένα κέντρο, σημείο μάλλον καινοτομίας, τα πιο καινοτόμα αποτελέσματα τα είχαμε με μια διατομιακή προσέγγιση. Για παράδειγμα, είχαμε μια συνεργασία ανάμεσα στην βιομηχανία αεροσκαφών και ε, τη βιομηχανία, την ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Είχαμε σπουδαία αποτελέσματα, πιο συγκεκριμένα η συνεργασία μείωσε τον χρόνο ανάπτυξης από τα τρία έτη στα ένα. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσίαση του προϊόντος τους, προϊόντος τους γίνεται ε, πολύ πιο ε, αποδοτική. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν όλα αυτά. Αυτή είναι η δική μου προσωπική εμπειρία ε, επιτόπου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στην κυρία Αΐντα Κατάνα από μια ε, εταιρεία συμβούλων στην ε, Ρουμανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με τα γενικά σχόλια, τα οποία έχουν να κάνουν με το κλίμα μέσα στο οποίο ετοιμάσαμε αυτή την παρουσίαση. Εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό συμμετέχω μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τις ε, δημόσιες υπηρεσίες και μέσω της διακρατικής συνεργασίας με την, ε, με την Βουλγαρία σε προγράμματα σαν αυτά τα οποία σας ε, παρουσίασαν οι συνάδελφοι προηγουμένω, αλλά και αυτά που θα σας δείξω εγώ. Παίρναμε στην επόμενη διαφάνεια. Ο κύριος Υπουργός που ήταν εδώ μαζί μας μας έλεγε πως έχουμε κοινέ υποδομές, ε, κοινέ στα δύο κράτη και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία προσπαθούμε να τις ε, ενισχύσουμε Άρα λοιπόν οι υποδομές είναι ένας κλάδος στον οποίο εργαζόμαστε και στις δύο χώρες και κυρίως για project τα οποία γίνονται στις ακτές του Δούναβη, στις όχθες του Δούναβη. Ένα ακόμα project το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αυτό της αλλαγής της συμπεριφοράς του πληθυσμού. Τι σημαίνει καινοτομία. Σημαίνει νέες εταιρικές σχέσεις πολύ γρήγορα. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Τι έχουμε εδώ. Στην περίπτωση των νέων κρατών μελών, ε, πρέπει να πω πως έλαβαν πάρα πολλά κονδύλια για να βελτιώσουν τις υποδομές τους και κυρίως το χώρο των μεταφορών. Πρέπει να σας πω ότι και στο παρόν και στο μέλλον τα νέα κράτη-μέλη που θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα διαφορετικά ταμεία θα το κάνουν. Σίγουρα ε, όμως θα μπορούσαν να στοιχηματίσουν και υπέρ της καινοτομίας γιατί όταν κάποιος αξιολογητής ή εκτιμητής αποφασίζει αν αξίζει η χρηματοδότηση ένα project ή όχι λαμβάνει υπόψη το κατά πόσο έχει παρουσιάζει κάποια καινοτόμα στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το project μπορούμε να στηρίξουμε την καινοτομία. Όλα αυτά με οδηγούν στο εξή συμπερασμά. Βεβαίω η καινοτομία μπορεί να ενταχθεί σε οποιοδήποτε project, είτε ε, αμυγός χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε συγχρηματοδοτούμενο και από τι εθνικέ κυβερνήσεις. Και βέβαια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να στηριχθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τι εθνικέ κυβερνήσεις γιατί προσφέρουν υπηρεσίες τι πάντα μπορούν να βελτιώσουν μέσω τη καινοτομία. Επόμενη διαφάνεια. Ξεκινώ εδώ κάνοντας μία ανάλυση των βασικών αξώνων που έχουμε στα κλαδικά προγράμματα και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, αλλά και σε κάποια από τα άλλα κράτη, νέα κράτη-μέλη. Μιλάμε εδώ για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος. Πολλά χρήματα έχουν διατεθεί μέσω μιας εταιρική σχέσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και εθνικής κυβέρνησης. Πολλές έχουν χρηματοδοτήσει έρευνες στα πανεπιστήμια και στα Ινστιτούτα Τεχνολογίας. Όμως πρέπει να δούμε γιατί δεν είναι αποδοτικά. Να σας πω το εξή. Η απορρόφηση, για παράδειγμα, είναι πολύ χαμηλή. Πρώτον, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν έχουμε πολλές αιτήσει. Και δεύτερον, υπάρχει μια μειωμένη δυνατότητα διοργάνωση τέτοιου είδων εταιρικών σχέσεων από όλες τις πλευρές. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια σχέση που θα μα πάει μέχρι τα μισά του δρόμου, δηλαδή κάποια projects τα οποία θα μπορέσουμε να εντάξουμε ε, και όσους έχουν πείρα από τέτοια προγράμματα για να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία τους και να προωθήσουμε τα προγράμματά τους. Εάν λοιπόν τονίζαμε περισσότερο την παρουσίαση των προτεραιοτήτων που έχουμε στα επιχειρησιακά προγράμματα και για να ξεπεράσουμε τις ε, συμφορήσεις που, που δημιουργούνται, τότε δεν θα είχαμε πρόβλημα. Σε περιφερειακό όμως επίπεδο θα πρέπει να έχουμε περιφερειακές στρατηγικές κοινοτόμες για να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Να δούμε όμως ποιος είναι ο κύριος αυτής της ε, στρατηγικής, γιατί εμείς δεν έχουμε τις απαραίτητες ε, δομές και τα αρμόδια τμήματα στις χώρες μας. Άρα λοιπόν τα διάφορα περιφερειακά συμβούλια δεν τα καταφέρουν αρκετά και στα όσα κάνουν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουμε την απαραίτητη συνεισφορά των εμπειρογνωμών. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια που είναι σχετική με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται αυτή τη ε, προγραμματική περίοδο η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Βλέπουμε λοιπόν πως δεν έχουμε απορρόφηση των κονδυλίων στη Ρουμανία. Αυτό αποτελεί πραγματικό πρόβλημα, γιατί κάποιες δεν επιβίωσαν τις κρίσεις και κάποιες άλλες, παρόλο που προσπάθησαν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, ετήθηκαν χρηματοδότηση, δεν μπορούν να αναλάβουν το τμήμα της ίδιας χρηματοδότησης. Εκεί λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταλάβουν πως χρειαζόμαστε μία ακόμα σπρώξια, έτσι ώστε αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να παρουσιάσουν project στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να το κάνουν και βέβαια να τεκμηριώσουν κάπως το ότι μπορούν να εξασφαλίσουν αντιμετωπίζουν την πτυχή καινοτομία. Χρειαζόμαστε κοινού κανόνε αξιολόγηση. Ε, για την επόμενη διαφάνεια, να δούμε τι, σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε. O altă problemă cred că se referă la capacitatea companiilor mici și mijlocii de a ένα ακόμα πρόβλημα είναι το κατά πόσο μπορούν να συνάψουν εταιρικέ σχέσει με τους ακαδημαϊκούς κύκλους, με τα πανεπιστήμια και με τοπική αυτοδιοίκηση, όπω σα είπα και προηγουμένω. Παρόλο που σε επίπεδο δηλώσεων και λόγων ή ε, προγραμματικών ε, δηλώσεων βεβαίως αποδίδεται προτεραιότητα στην ε, συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού κλάδου και πανεπιστημίων, στην πραγματικότητα συμβαίνει ελάχιστα. Και επιπλέον πολλές φορές οι οι επιχειρήσεις δεν έχουν μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη στρατηγική και δεν βρίσκουν ε, τι μέλλον θα έχει αυτή η εταιρική σχέση με τα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει λόγος να το εφαρμόσουν, ούτε καν με κέντρα ερευνητικά, γιατί πολλές φορές τα αποτελέσματα τα βλέπει κανείς μετά από πέντε χρόνια. Μια πενταετία. Τι να γίνει λοιπόν όταν η μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει τόσο μακρόπνοα σχέδια. Ακαδημαϊκοί κύκλη. Τα κέντρα τα ερευνητικά πολύ σπάνια δέχονται να συνεργαστούν με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Συνήθως η έρευνα θεωρείται ως κάτι που ωφελεί την ανθρωπότητα, αλλά όχι το άτομο. Έτσι λοιπόν για τους ακαδημαϊκούς κύκλους πιστεύω ότι θα πρέπει οι, εκεί να λάβουν υπόψη την πτυχή άνθρωπος, άτομο, κοινότητα και να βρούνε πιο γρήγορα μια κοινή γλώσσα και έναν τόπο τομής. Το 2003 όταν Κοίταξα να δω πώς χρησιμοποιούνται στην στα Midlands στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια. Είδα πως ε, είχαμε συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών κύκλων τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού ε, κλάδου, ε, συνεργασία πολύ στενή που βασιζόταν σε μια πολύ ξεκάθαρη βάση ε, εταιρικής σχέσης με αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη αυτήν την κουλτούρα της εταιρικής σχέσης και της καινοτομίας να την αναπτύξουν. Τότε μόνο θα βελτιωνόταν τα πράγματα και θα είχαμε καλύτερη χρήση απορρόφηση και αποδοτικότητα των ε, σχετικών ε, ταμείων. Να λοιπόν τα καυτά σημεία τα μπορούμε να εντοπίσουμε στην διαδικασία διαχείρισης των project, το management. Τα βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια. Προγραμματισμός, ε, ορισμός και αξιολόγηση. Διαφορετικά δεν έχουμε ένα πλαίσιο αναφοράς. Εάν λοιπόν δεν έχουν μακρομεσοπρόθεσμη στρατηγική μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς θα καταφέρουμε να πάρουμε κάτι το οποίο να έχει πραγματικό αντίκτυπο. Διαφορετικά ζούμε σε σφαίρες πολύ μακριά τη πραγματικότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να ε, οριστεί με λεπτομέρειε το project και μετά βεβαίως να αξιολογηθεί η πτυχή της καινοτομία, έτσι ώστε η εκχώρηση κοινοτικών κονδυλίων να γίνει, γιατί θα είναι γνωστό πού οδηγεί αυτό το project και τι προσφέρει σε επίπεδο καινοτομία. Αξιολόγηση λοιπόν των προτάσεων που υποβάλλονται με, μεθοδολογία η οποία είναι τυποποιημένη και με του απαραίτητου πόρου, του ανθρώπινου, για να γίνει η αξιολόγηση τη καινοτομία που προσφέρει αυτό το project. Σε επόμενε δύο διαφάνειε παρουσιάζω κάποια παραδείγματα για να δούμε τι έχει γίνει. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε στο περιφερειακό επιχειρησικό πρόγραμμα της Ρουμανίας το κριτήριο για την κοινωνία της πληροφορίας και της νέες τεχνολογίες. Εδώ, στην καινοτομία, δίνουμε έξι βαθμούς. Έξι από τους εκατό που θα μπορούσαμε να δώσουμε όλα αυτά το κριτήριο είναι γνωστό, δηλαδή τεχνολογία της κοινωνίας της πληροφορίας. Θα έπρεπε να έχει υψηλότερη βαθμολογία. Μετά έχουμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που το αποδεικνύει. Εννέα, εννέα βαθμούς παίρνει κανείς εκεί για την καινοτομία από ένα σύνολο 100 βαθμών που μπορεί να δοθεί σε ένα συγκεκριμένο project για να προκριθεί. Αυτά λοιπόν που είπα προηγουμένως θα τα συνοψίσω εδώ στα συμπεράσματα. Καταρχήν, στο στάδιο του προγραμματισμού, εάν γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων περιφερειακών και τοπικών φορέων, θα έδινε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό βέβαια ισχύει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα εθνικό πλαίσιο αναφοράς που να αναφέρεται στην καινοτομία και που να παραπέμπει στους κλάδους όπου η τεχνολογία και η έρευνα θα δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Δομημένη πληροφορία που θα δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί εάν δεν δίνονται με διαρθρωμένο τρόπο, δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητές και δεν είναι εύληπτες. Μεθοδολογία και κοινοί κανόνες, κοινή μεθοδολογία. Αυτό μας είπε και ο Υπουργός της Βουλγαρίας. Οι δήμαρχοι πρέπει να βλέπουν μία σαφή μεθοδολογία στις προτάσεις που κατατίθενται και θα πρέπει να έχουν κατευθυντήριες γραμμές για να ξέρουν πώς θα δράσουν. Αυτή είναι μια κοινή ανάγκη και βέβαια θα πρέπει να προωθήσουμε ε, project τα οποία θα προωθήσουν την κουλτούρα τη συνεργασία, τη εταιρική σχέση. Να δούμε τι γίνεται στη Ρουμανία και στα άλλα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να κάνουμε καινοτομία χωρί να υπάρχει πραγματική συνεργασία. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Η πρόεδρος Ιπνερ. Τελευταίος ο κύριος Χέλμουτ Γέγκερ Είσαστε από το... Έχει τέλο πάντων την τελευταία ομιλία. Θα μας αναπτύξετε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πρώτα πολύ για την πρόσκληση. Το Braunschweig βρίσκεται στα σύνορα της γραμμής που χώριζε τις δύο Γερμανίες. Έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα ερευνητικών κέντρων θα σας εξηγήσω πώς αρχίσαμε το 1982 με την τεχνολογία της ηλιακής ενέργειας, στην αρχή για πισίνες, μετά για το ζεστό νερό. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 ε, προχωρήσαμε στην θέρμανση με ηλιακή ενέργεια. Το 2002 φτιάξαμε ένα κτίριο εργοστασίου με μηδέν εκπομπές αερίων που υποστηρίχθηκε και από και κοινοτικά ε, ταμεία κατά 10,5%. Έχουμε εδώ τις δραστηριότητες μας οι οποίες έχουν βραβευθεί. Δεν θα σας τις αναπτύξω. Αν θέλετε παρακαλώ προχωρήστε στην επόμενη διαφάνεια. Η παλέτα των προγραμμάτων μας περιλαμβάνει θερμάνσεις, ηλιακούς συσσωρευτές, τους σχετικούς ρυθμιστές, επίσης ε, εγκαταστάσεις θερμάνσεως για πολυκατοικίες, για ξενοδοχεία, για νοσοκομεία, φωτοβολταϊκά συστήματα και το καθεξής. Από την βιοτεχνική αυτή πρώτη ανάπτυξη έχουμε προχωρήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών που μπορούν να θεωρηθούν υψηλής τεχνολογίας, high tech. Εδώ βλέπετε κατά ε, εγκατάσταση συγκολήσεω χαλκού και αλουμινίου. Νέα τεχνολογία αυτή που ε, στην Γερμανία μας έχει επιτρέψει να κατακτήσουμε 30,5% της αγοράς ε, για τις για τα συστατικά αυτά ε, συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται σε ε, ηλεκτρικούς ε, σε ηλιακούς μάλλον συλλέκτες και μπορέσαμε να μειώσουμε το κόστος κατά 20% περίπου. Επόμενη διαφάνεια, το κύριο βάρος των δραστηριοτήτων μας είναι η ένταξη της ηλιακής τεχνολογίας στα συστήματα θερμάνσεως. Αυτή είναι και η καινοτομία για μας ε, που αναπτύξαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή στα συστήματά μας πρώτη στο ρόλο παίζει ο ήλιος και όταν δεν επαρκεί το ηλιακό φως τότε ε, μπαίνει σε λειτουργία πλέον είτε το πετρέλαιο είτε το φυσικό αέριο είτε οι αντλίες θερμότητος που ε, χρησιμοποιούν την θέρμανση του εδάφους. Για τις καινοτόμες αυτές τεχνολογίες έχουμε λάβει πολλές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια της International Energy Agency συμμετέσχομεν σε ένα τεστ ε, συγκρίσεως και αποδείχθηκε ότι το σύστημά μας είναι από τα πλέον αποτελεσματικά, τα πλέον αποδοτικά. Βλέπετε τώρα την πιο πρόσφατη ε, εξέλιξη της ε, επιχειρησεώς μας, μια αυτόματη ε, εγκατάσταση που έχει συνολική έκταση 2.000 τετραγωνικά μέτρα με την αυτοματοποίηση αυτή μπορέσαμε να μειώσουμε το κόστος χρήσεως κατά 30% και με την τεχνολογία αυτή είμαστε σε θέση να παράγουμε στο Braunschweig σε ανταγωνιστικές τιμές επίπεδους συλλεκτήρες. Βλέπετε πάλι εδώ ε, κάποιες απόψεις του κτηρίου μας, το οποίο όπως είπα έχει μηδενικές εκπομπές, για να μπορούμε να δείξουμε και στους πελάτες μας τι μπορούμε να επιτύχουμε με, με τη σύγχρονη αυτή τεχνολογία. Έχουμε περίπου χίλιους ε, ιδιωτικούς επισκέπτες και πάνω από χίλιους ε, ε, βιοτέχνες οι οποίοι έρχονται και μας επισκέπτονται. Βλέπετε εδώ ένα τυπικό παράδειγμα στη Γερμανία, μια μονοκατοικία κοντά στην πόλη Ανόβερο. Βλέπετε ότι το σπίτι με την παλαιά τεχνολογία που χρησιμοποιούσε, χρησιμοποιούσε και 2.250 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Με, την αντικατέστησε αυτή και έχει κατεβάσει την ε, κατανάλωσή του στα 1.200 κυβικά μέτρα ε, φυσικού αερίου. Παρακαλώ η επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ την ροή της ενέργειας στα πλαίσια του εργοστασίου μας. Εμείς χρησιμοποιούμε μόνο εναλλακτικέ ε, πηγές ενέργειας, 20% από φωτοβολταϊκά έργα, ε, αλλά προέρχονται από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας τα οποία κάνουν συμπαραγωγή ενέργειας. Το, όλο το κτίριό μας έχει ε, συστήματα ανάκτησης της ενέργειας, δηλαδή η θερμότητα η οποία θα εκλειόταν απλώς στον αέρα ε, επανακτάται και μάλιστα εγκαταστήσαμε ένα σύστημα απορρόφησης του, του ψύχους με το οποίο μπορούμε είτε να θερμαίνουμε είτε να ψύχουμε το εργοστάσιό μας λόγω με την ε, εποχή. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα ίχνος ενέργειας που να μην επαναχρησιμοποιείται με αποτέλεσμα βέβαια η εξοικονόμηση της ενέργειας να είναι τεράστια. Βλέπετε εδώ μια εικόνα του εργοστασίου μας που το 2002, 2002 ε, συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικέ πηγές σε τάξη του 7,5%. 90% των ερευνητικών μας προγραμμάτων χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους, 10 περίπου των ε, ε, ερευνών μας έγιναν με κοινοτική χρηματοδότηση κάτι το οποίο κατέστη δυνατόν μόνον διότι ορισμένα Ινστιτούτα όπως το Fraunhofer ή άλλο Αυστριακό Ινστιτούτο ανέλαβαν την, τον συντονισμό των ε, ερευνητικών αυτών προγραμμάτων. Εμείς ως μικρή επιχειρήση δεν ήμασταν σε θέση να ζητήσουμε και να επιτύχουμε ε, κοινοτική χρηματοδότηση. Τώρα η εικόνα του 2008 όπου το 2008 μπορέσαμε και διπλασιάσαμε στα 15.000 τετραγωνικά μέτρα την έκταση του εργοστασίου μας. Παράγουμε συστήματα υψηλής τεχνολογίας για την ε, θέρμανση, κυρίως για μεγάλα κτίρια όπως νοσοκομεία αλλά και πολυκατοικίες. Ποιες ήταν οι εμπειρίες μας τα τελευταία 10 χρόνια με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να βελτιωθεί λίγα σχόλια ακόμη για το τέλος της ομιλίας μου. Τα συμβουλευτικά γραφεία για τις κοινοτικέ χρηματοδοτήσεις στη Γερμανία εν τω μεταξύ γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα. Υπάρχουν και φίρμες παροχής συμβουλών που είναι πάρα πολύ ικανές. Το μέγα πρόβλημα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ο συντονισμός με άλλους εταίρους. Όταν δηλαδή πρόκειται να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα όπου πρέπει να συμμετέχουν τρεις ή τέσσερις χώρες, υπάρχουν ε, μακροχρόνιες συζητήσεις για ε, την εκμετάλλευση ε, του αποτελέσματος της έρευνας και η πρότασή μας θα ήταν στο μέλλον ίσως να δίνεται η δυνατότητα να ζητούν και εταίροι από δύο μόνο χώρες ε, τη χρηματοδότηση αυτή, ώστε να ε, συλλέγουν εμπειρίες σε μια πρώτη φάση για να μπορέσουν μετά να συνεργαστούν και με περισσότερου εταίρους. Το μέγα πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι η, μακρύ, η, μακρά διάρκεια του χρόνου επεξεργασίας των αιτήσεων. Γίνονται μεν αναέτος οι προκηρύξεις, μετά από τι προκηρύξεις κατατίθενται ε, οι προτάσεις έργων, αλλά συχνά περνούν μέχρι και 9 μήνες μέχρι ότου ε, ληφθούν οι χρηματοδοτήσεις. Αλλά για μια μικρομεσαία επιχείρηση ο χρόνος αυτός είναι πάρα πολύ μακρύς, διότι όταν μια μικρομεσαία επιχείρηση έχει ε, μια ιδέα, καινοτόμο ιδέα, την ενδιαφέρει το ταχύτερο δυνατό να την προσφέρει στην αγορά. Αυτές, αυτοί οι χρόνοι λοιπόν πρέπει να συντομευθούν. Οι εμπειρίες μας είναι επίσης ότι η κοινοτική χρηματοδότηση απευθύνεται κυρίως σε μεγάλα έργα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σαφώς άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ που για τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ουσία είναι αδύνατον να συγχρηματοδοτήσουν κατά το αντίστοιχο μέρος για αυτές ε, έργα τέτοιου ε, ύψους. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που κάνατε. Μια παρουσία. Ε, ήταν μάλιστα εισηγήσει οι οποίε ήταν ε, παραπληρωματικέ, γιατί, γιατί όλοι σα ε, τονίσατε διάφορε πτυχέ αυτή τη διαδικασία που είναι η καινοτομία και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσει και να κάνουν σχόλια. Ο Σον Κέλλη είναι ο πρώτο. Καταρχήν, Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπαν. Ίσως και πάρα πολλά για να τα απορροφήσει κανείς και να θυμηθεί όλες τις ε, λεπτομέρειες. Ξεκινάω με τον Τζον Μάλς που είναι και συμπατριώτης μου. Ανέφερες ότι 12,2 δεις πάνε στι καινούργιες εταιρείε. Πόσες από αυτές θεωρείς ότι είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Δεύτερη ερώτηση, ανέφερε στη διαφορετική ένταση. Όμως νομίζω πως η, Ιρλανδία είναι κάτω-κάτω στη σειρά. Αλλά και η Γαλλία. Υπάρχουν ειδικοί λόγοι γι' αυτό. Μίλωσες επίσης για ε, λανθάνοντες καινοτόμους τι θα κάνουμε για να τους ξυπνήσουμε και να τους βρούμε. Ο κύριος ε, Νίσενς νομίζω είπε ότι χρειάζεται η αλλαγή από την νοοτροπία της στήριξης στην στρατηγική την, ε, στήριξη μάλλον προγραμμάτων, στη στήριξη περιφερειακής στρατηγικής. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτρης Σίμων, παρακαλώ. Επιτέλους. Το είπα με γερμανική προφορά το όνομά σα. Σα ευχαριστώ. Κάνει ένα πρόβλημα. Έχοντας ακούσει την τελευταία παρουσίαση σχετικά με την δυσκολία να εγκριθούν τέτοια έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή είναι θέμα μεγάλης χρηματοδότησης. Αυτό συμφωνεί και με την εμπειρία από εθνικά προγράμματα που εμπίπτουν στο, στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας. Η καινοτομία για πολλούς προέρχεται από επιχειρήσεις οι οποίες συχνά ήταν πολύ, εγκατισμένες πολύ μακριά για χρηματοδοτήσεις από τα τρέχοντα διαθωτικά ταμεία για το λεγόμενο cluster management σε όλη την αλυσίδα δημιουργίας αξίας που θα επιτρέψει στους μεγάλους παίκτες της βιομηχανίας οι οποίοι ούτως ή άλλως ασχολούνται με την καινοτομία να συνδυάσουν τις προσπαθειές τους και με τους μικρούς οι οποίοι βρίσκονται σε τελείω διαφορετική μεριά ή μπορεί όμως να παίζουν το ρόλο του προμηθευτού ή θα υποφεληθούν από το προϊόν τελικά της βιομηχανικής παραγωγής και μέσα σε αυτό το κλάστερ να υπάρξουν ροές καινοτομία από τους μεγάλους προς τους μικρούς. Αυτά είναι δυνατά τώρα, τέτοιοι συνδυασμοί δηλαδή. Δεν έχουμε όμως ακόμα επιτυχίες, να πούμε δηλαδή ότι ναι, πράγματι τέτοιο ποσοστό επιτυχίας. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι, θα, πείτε, θα, θα, δεχτείτε ότι είναι επιτυχημένη η στρατηγική αυτή να προχωρήσουμε δηλαδή σε υποστήριξη από τα λεγόμενα κλάστερ, τα κέντρα διασποράς, δηλαδή με συνδυασμό προσπαθειών επιχειρήσεων μεγάλων με μικρές ή νομίζετε ότι πρέπει να γίνει μονάχα μέσα σε συγκεκριμένους τομείς. Μία ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Ένα ακόμα σχόλιο από τη Φραντζέσκα Ντε Τον, συγγνώμη, ε, ευχαριστώ. Εγώ άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει να πω ότι ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσε οι εισηγήσει. Θέλω να θα απλοποιήσω γιατί δεν υπάρχει χρόνο για να εμβαθύνουμε. Είναι τεράστια συμμαχία η πολιτική συνοχή. Δηλαδή η σχέση με τι μικρομεσαίες επιχειρήσει που αντιπροσωπεύουν την ράχο κοκαλιά τη οικονομία μα. Ε, come favorire Πώς μπορούμε να ευνοήσουμε τη διαδικασία ολοκλήρωσης ε, και μάλλον σώρευσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, πράγμα το οποίο θα καταστήσει πιο στεναρό, πιο στέρεο τον ιστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έπειτα, η απλοποίηση και η επιτάχυση των διαδικασιών ε, των δαπανών ε, της χορήγησης των κονδυλίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη διάφορα προβλήματα. Προβλήματα πρόσβασης στις πιστώσεις, προβλήματα ρευστότητας. Σε μια κατάσταση κρίσης πραγματικά κινδυνεύουν να πτωχεύσουν. Το θέμα λοιπόν του χρόνου είναι ουσιαστικό, είναι προτεραιότητας. Άρα, ποια μέσα θα πρέπει να απλοποιήσουμε και να ε, επιταχύνουμε. Τρίτο ερώτημα. Πώς να βρούμε και να αφυπνίσουμε τους ε, λανθάνοντες καινοτόμους. Πώ θα χτυπήσει αυτό το ξυπνητήρι έτσι ώστε αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να συμβαδίσουν με τα καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα. Τελευταία ερώτηση και κλείνω. Όσον αφορά τους, τα κέντρα καινοτομίας και αριστείας. Ε, αυτό είναι ο στόχος, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να είναι ανταγωνιστικές για να μπορούν να σταθούν στην αγορά και να ξεπεράσουν την δύσκολη πρόκληση της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει ακριβώς επειδή είναι μικρές και πολύ συχνά ακόμη πιο μικρές από μικρές ε, να βασιστούν στην καινοτομία, στην αριστεία, στο know-how που θεωρώ ότι είναι το χαρτί που μπορεί να επιτρέψει στην ενίσχυση του ιστού στην Ευρώπη των μικρών, των πολύ μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τους εισηγητές να απαντήσουν. Φυσικά μπορείτε να σχολιάσετε και στοιχεία τα οποία, ε, ερωτήσεις που δεν, ήταν, δεν απευθύνθηκαν σε εσάς, αλλά που θεωρείτε ότι, μπορείτε, ε, ότι έχετε κάποια άποψη να πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω λοιπόν ακούσει κάποιες ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσω άμεσα και θα ε, σχολιάσω και κάποια από τα υπόλοιπα. Οι εταιρείε που ξεκινάνε σήμερα, οι μικρομεσίες αυτές, τα startup, είναι βιώσιμα. Κοιτάξτε, η επιλογή project ε, σε αυτό το χώρο είναι από τις διαδικασίες που πιο πολύ καθυστερούν Άρα λοιπόν βλέπουμε πως τέτοιου είδους στήριξη είναι αυτή που μας λιγότερο που μας ζητάνε λιγότερο και όπου οι επιδόσεις μας είναι πολύ αργές. Δεν είναι πολλές οι εταιρείε ή τα άτομα τα οποία σε αυτή την τρέχουσα συγκυρία ξεκινάνε μια δικιά τους επιχείρηση. Μην ξεχνάτε όμως πως εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρουμε αν είναι βιώσιμες ή όχι, γιατί έχουν επιλεγεί από οι υπηρεσίε σαν αυτή της Δυτικής Ολλανδίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οπότε εκείνοι κρίνουν για το ποια είναι τα πιο ενδεδειγμένα μέτρα και παρόλο που αυτά τα startup είναι μια ομάδα που καθυστερεί, αυτό που είδαμε ήταν μια στήριξη του δανειακού κεφαλαίου έτσι ώστε να στηριχθούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις αυτή την εποχή της κρίσης. Πολύ καλή ερώτηση όμως και είμαι σίγουρη πως οι ε, διαχειριστικές αρχές και οι αναπτυξιακές εταιρείες κάνουν, ε, παίρνουν κάποιες αποφάσεις δύσκολες στη στιγμή της επιλογής. Εμείς τουλάχιστον στο δικό μας επίπεδο βλέπουμε πως η στήριξη για τις εταιρείες αυτές, τις καινούριες, τα start-up, δεν τρέχει με τους ρυθμούς που θα θέλαμε και μάλλον αυτό οφείλεται στην κρίση. Για τη διαφορά σε επίπεδο στήριξη της μικρόμεσες επιχειρήσεις, η Ιρλανδία όντως βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις, όπως ε, μας είπε ο συνάδελφός σας, γιατί βέβαια από την περίοδο 2000-2006 στη νέα προγραμματική περίοδο εκεί η επιλογή της Ιρλανδίας ήταν να εστιάσει σε άλλες προτεραιότητες στα δύο περιφερειακά προγράμματα και να αφήσει στην άκρη την επιχειρηματική στήριξη. Άρα λοιπόν είναι ασυνήθιστα χαμηλή η χρήση των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έχουν όμως πολύ υψηλά κονδύλια εθνικής προέλευσης και πολύ καλή πολύ καλά παραδείγματα από το παρελθόν στη στήριξη επιχειρήσεων. Στη Γαλλία όπως και σε κάποια άλλα κρατημέλη, η μέση στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα είναι στο 10% αντιπροσωπευτικό του τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στην σύγκληση, μια και η ε, Γαλλία είναι ανταγωνιστική, τουλάχιστον η υπηρετική ε, Γαλλία δεν είναι χώρα σύγκλησης, έχουν ε, δώσει την προσοχή τους στις διάφορες κατηγορίες από τη Λισαβόνα και νομίζω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στα πλαίσια του earmarking που γίνεται για την ατζέντα της Λισαβόνας. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούν πως η στήριξη επιχειρήσεων είναι κάτι μεμονωμένο που στηρίζει μόνο κάποιες επιχειρήσεις. Εμείς όμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και αρκετά χρόνια στηρίζουμε μια πιο περιφερειακή προσέγγιση. Και η πιο πρόσφατη προσπάθεια είναι μια κοινή ανακοίνωση όλων των εμπλεκόμενων επιτρόπων για την περιφερειακή πολιτική και την ευφύ ανάπτυξη, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ευφυή εξειδίκευση αυτή τη στρατηγική και ο κύριε Νίσκενς νομίζω πως και χωρίς την ευρωπαϊκή στήριξη μπορεί να θεωρηθεί τόσο ένα εξαιρετικό παράδειγμα στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης. Τώρα για τόσα είπε η κυρία Κατάνα, Πιστεύω πως η μελέτη στην οποία αναφέρθηκα για την αξιολόγηση της καινοτομίας και τη στήριξη καινοτομία έχει και κάποια εθνικά κεφάλαια. Και τα αποτελέσματα μπορείτε να διαπιστώσετε από το τι συνέβη στα άλλα κράτη-μέλη, από την αξιολόγηση εκεί των μέτρων στήριξης και αξιολόγηση. Ίσως λοιπόν από τα άλλα κράτη να βρούμε κάποια διδάγματα και εμπειρίες που να μπορέσουμε μετά να ανταλλάξουμε επιτυχώς. Το τελευταίο που έχω να πω είναι πως σε σχέση με τις συνέργειες ή την έλλειψη συνέργειας που διαπιστώνεται μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σας πω πως έχουμε ένα πολύ δημοφιλές εγχειρίδιο, έναν οδηγό για τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα. Είναι ένα διαδραστικό site σε όλες τις επίσημες γλώσσες έτσι νομίζω, και βρίσκεται στον ισότοπο κόρτης. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύχριστο και χρήσιμο εργαλείο ε, για να γνωρίσει καλύτερα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα και βέβαια αυτό συμπεριλαμβάνει και την κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποια σχόλια για αυτή την αλλαγή πολιτικής από τα μεμονωμένα project σε μια πιο περιφερειακή προσέγγιση στήριξης. Η περιφερειακή αυτή προσέγγιση σημαίνει ότι όλα τα χρήματα μπαίνουν σε ένα καλάθι, δηλαδή στηρίζουν μία πολιτική. Και βέβαια όταν κανείς ε, το οργανώσει καλά η περιφέρεια είναι ε, ικανή να επιλέξει τους κλάδους που έχετε τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας για το μέλλον, όπου θα γίνεται στο μέλλον πιο ανταγωνιστική. Όταν λοιπόν έχετε τέτοιου είδους συνεργασία, τότε οι παίκτες έρχονται σε εσά άμεσα από τις επιχειρήσεις, από τις κυβερνήσεις και στέκονται δίπλα σας. Το οποίο σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά κάθε χρονιά. Όταν μιλάμε λοιπόν για ταμείο συνοχή και όταν μιλάμε για μετακίνηση από την μεμονωμένη στήριξη στην περιφερειακή στήριξη, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, στηρίζεις μια γενικότερη κατεύθυνση και αυτό ισχυροποιείται από τη συμβολή των υπολείπων. Τώρα, για το sleeping innovation, ε, όταν έχουμε μια τέτοια προσέγγιση εχμής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να όπως όλα συνηγορούν έτσι ώστε οι προσπάθειες που κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ευθυγραμμιστούν Μπορεί λοιπόν να είναι κανείς σε επαφή με μικρομεσαίες με τις οποίες δεν μπορεί να βρεθεί κανείς αλλού να συναντηθεί. Αυτό είναι το πλεονέκτημα στις προσέγγισης. Έρχεσαι σε επαφή με επιχειρήσεις γιατί είναι σε κάποιο δίκτυο ή γιατί συνεργάζονται μεταξύ τους. Στην πράξη λοιπόν αυτό προσφέρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. γιατί βέβαια έχουμε και την εγκάρσια διακλαδική προσέγγιση ε, που και αυτή δεν είναι τόσο συχνή. Πάντως συνήθως οι επιχειρήσεις περιοριστούν στη δική τους αλυσίδα στις προσπάθειες που κάνουν και αυτό πρέπει εσείς να τους οργανώσετε έτσι ώστε να ακολουθήσουν μια διακλαδική προσέγγιση. Στον κλάδο της συντήρησης έχετε τις διάφορες επιχειρήσεις, ε, τη μεταποιητική, τον κλάδο της ενέργειας, τον κλάδο των υποδομών, έχετε τον κλάδο της αεροναυπηγικής. Θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί να συνεργαστούν με επιχειρήσεις τις οποίες δεν γνωρίζουν. Έτσι όμως επιταχύνεται η διαδικασία της καινοτομίας και γνωρίζετε πως έτσι μπορείτε να βρείτε και αυτού του sleeping innovators, του οποίου διαφορετικά δεν θα βρίσκατε. Θα ήθελα να απαντήσω στα όσα είπαν ο κύριος Ντεάντζελης και ο κύριος Κέλλη για το πώς μπορούμε αυτούς τους sleeping innovators με αυτούς τους sleeping innovators και το τι έγινε με τη συμφωνία μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας. Έχουμε ένα σχέδιο εντοπισμού και αν δω την περιοχή Γον Αλπ, είχαμε τους ενδιάμεσους που ήταν τα εμπορικά επιμελητήρια και ε, τις ε, επαγγελματικές οργανώσεις όπου οι περιφέρειες χρηματοδότησαν συμβούλους από αυτές τις οργανώσεις που πήγαν επί τόπου, συναντήθηκαν με τις επιχειρήσεις και βρήκανε 50 ε, υπνώτες κάθε χρόνο και ε, αυτοί τους βοήθησαν να βρουν άλλους 50 κάθε χρόνο. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν περιοχές τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Μιλάμε για 100.000 τέτοιες περιπτώσεις που ανιχνεύτηκαν σε τρεις μόνο περιοχές. Δεύτερη και τρίτο παράδειγμα μάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να σας πω πως είναι συνήθως αυτή η κόμβη ε, περιφερειακής καινοτομίας που ευαισθητοποιούν όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, έχουμε μαθήματα επιμορφωτικά, τα οποία προσφέρουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι βιοτεχνικές οργανώσεις, τα επιμελητήρια ε, κάθε κλάδου που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων και σπουδών για θέματα προσαρμογής στις νέες και καινοτομίας, και δίνουν παραδείγματα καινοτομία που έγινε από τις αντίστοιχες εταιρείε. Γιατί η μικρομεσαία επιχείρηση αυτού του είδους τα μαθήματα είναι πολύ σημαντικά. Το να βρει κανείς λοιπόν αυτούς που φέρουν την καινοτομία γίνεται, γίνεται σε διάφορες περιφέρειες και αυτό που χρειάζεται είναι μια εκστρατεία πανευρωπαϊκή για να δούμε πώς μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Μία προσθήκη για αυτό το θέμα και εγώ. Μήπως θα μπορούσαμε και για την κουλτούρα της καινοτομίας και της εταιρική σχέσης να κάνουμε κάτι παρόμοιο, να ευαισθητοποιηθούν και να γνωρίζουμε και εμείς πώς ασχολούνται με την καινοτομία. Ευχαριστώ να απαντήσω αφενός για τα κλάστα, τα ε, κέντρα ε, διασποράς και υπεροχής είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους για την πρόθεση της κοινοτομίας. Το πιο σημαντικό είναι οι μεγάλες εταιρείες που συμμετέχουν να είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με τις ΜΜΕ σε ισότιμη βάση. Γιατί συχνά οι ΜΜΕ έχουν πολύ συχνά τον φόβο ότι θα κλαπούν οι καινοτόμες ιδέες τους Άρα πρέπει να υπάρχει μια στέρεα βάση γιατί τελείως δεν θα είναι διατεθειμένε οι ΜΜΕ να συνεργαστούν. Πάντως, κατά τα άλλα, είναι θαυμάσια η δυνατότητα αυτή για την προώθηση των καινοτομιών, διότι ο, η μικρομεσαία επιχείρηση χρειάζεται σύντομου δρόμους. Αυτό κάνει και τόσο δύσκολες τις διαμεθοριακές συνεργασίε, διότι αν πρέπει ο επιχειρηματίας να καλύψει εκατοντάδες χιλιόμετρα για να πάει σε μια συνάντηση, δεν θα το κάνει τελικά. Άλλη σημαντική δυνατότητα εφαρμογής είναι σε όλα τα πανεπιστήμια να ανοίξουν κέντρα συμβουλών για την τεχνολογία, διότι και τα πανεπιστήμια και τα κέντρα ερευνών πρέπει να δραστηριοποιηθούν ώστε οι καινοτομίε που προωθούν να καταλήξουν στην αγορά. Η δεμή, οι περιφερειακές οργανώσεις ανάπτυξης μπορούν να αποδειχθούν επίσης ε, σημαντικοί παίκτες στην υπόθεση αυτή. Δηλαδή θα πρέπει να προσφέρουν πλήρη δυνατότητα παροχής συμβουλών για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Στο Braunschweig που είναι μια περιφέρεια η οποία επλήγει σοβαρά από την ε, από τις διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη δεκαετία του 90 και μέσα από την κρίση ξεκίνησε μια πρωτοβουλία με συμμετοχή ε, εργοδοτών και εργαζομένων ε, στην κατασκευή μηχανών που σήμερα, έχει τώρα, ε, που σήμερα συμμετέχουν σε αυτήν πάνω από 30 επιχειρήσεις και προωθεί και καινοτόμα project και που οργανώνει όμως ταυτόχρονα και από κοινού τις αγορές τις προμήθειες δηλαδή. Και έχει ε, αναπτυχθεί η παραγωγή στο πενταπλάσιο γιατί δεν ήταν ε, γνωστή και μέσα στην περιφέρεια τι προμήθευε ο κάθε προμηθευτής από τους μένους τους δε. Δέτοιες ε, οργανώσεις χρειαζόμαστε σε όλη την Ευρώπη. Κάτι άλλο που χρειαζόμαστε και που θεωρώ ότι θα είναι μια δύσκολη διαδικασία διότι απαιτεί μια αλλαγή νοοτροπίας γιατί αυτό θα ήταν βασικά καθήκον των ε, βιομηχανικών και εμπορικών επιμελητηρίων, που στην ουσία όμως αυτό που κάνουν είναι διαχειρίζονται το παρελθόν, αντί να ασχολούνται με την μελλοντική ανάπτυξη. Και ε, το επιμελητήριο του Braunschweig δηλαδή ασχολείται πολύ με τις πολιτικές επαφές στο Βερολίνο ή στις Βρυξέλλες, αντί να εγγύψει στα θέματα εκείνα στα οποία πραγματικά μπορεί να έχει ουσιαστική επιρροή. Γιατί ε, η, οικονομική ζωή του Σφάικ δεν έχει μεγάλη επιρροή στην πολιτική ζωή του Βερολίνου ή των Βρυξελών. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει το επιμελητήριο όμως θα ήταν να βοηθήσει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Χρειάζεται λοιπόν αλλαγή νοοτροπίας ή χρειάζεται εξειδίκευση, εξειδικευμένες μάλλον οργανώσεις ε, ανάπτυξης που θα επιληφθούν το θέματος και που θα έχουν μια άλλη νοοτροπία, πραγματικά καινοτόμο νοοτροπία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φανίστελρο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως μπορώ να είμαι σύντομος. Γιατί αν δούμε τα όσα μας παρουσιάστηκαν σήμερα εδώ, φαίνεται ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η περιφερειακή διάσταση της συνεργασίας. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στις περιφέρειες και άκουσα πολλούς να το λένε αυτό. Ορισμένοι λένε ποια είναι η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, αλλά Νομίζω πως σήμερα το βλέπουμε έμπρακτα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω πως ε, έχουμε δώσει αρκετή στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αν το κάνουμε αυτό έχουμε ηθαρρυντικά αποτελέσματα. Δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω και αυτό το απευθύνω στον κύριο Νάισκινς που είναι από την χώρα μου και από την περιφερειά μου. Ε, είπατε ότι δόθηκαν 592 εκατομμύρια ή όχι, 592.000 ευρώ, όχι, εκατομμύρια. Εκατομμύρια ήτανε. Αυτά επενδύθηκαν στην περιφέρεια. Θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν χωρί τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποια ήταν η προστιθέμενη αξία, τι πρόσθεσε η συμμετοχή της Ευρώπης, ε, ποια ήταν η σχέση ανάμεσα στην εμπλοκή της των Βρυξελών και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Ήταν αποτελεσματικός ο τρόπος. Συνεργασία, ο Γιάννου. Σας ευχαριστώ. Εγώ απευθύνομαι στον κύριο Τζον Watts βασικά. Αλλά ίσως και κάποιος άλλος από τους ομιλητές να θέλουν να απαντήσουν. Εμείς έχουμε συγκεντρώσει κάποιες αρχικές ε, εμπειρίες όσον αφορά την οικονομική μηχανική και λογιστική. Ε, έχω όμως κάποιες παρατηρήσεις. Τι, ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποια είναι τα συμπεράσματά της και πώς ετοιμάζεται για την επόμενη περίοδο. Γιατί στην εισήγησή σας διάβασα κάποιες τολμηρές προτάσεις όσον αφορά την αύξηση Μιλάτε για, όχι για επιδοτήσεις, αλλά για δάνεια, ε, ερευνητικές εγγυήσεις και ούτω καθεξής. Και εσείς πώς εκτιμάτε ότι θα γίνει δεκτό αυτό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί πρόκειται για μια πλήρη μετακίνηση από τις επιδοτήσεις στα δάνεια. Ποιε ήταν οι επιπτώσεις λοιπόν αυτού του νέου συστήματος και της εφαρμογής του, ποια ήταν η αντίδραση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ. Τυφλώθηκα ή ο Μάικλ Τόιερ, Μίκαελ Τόιερ δεν είναι πια στην αίθουσα. Μου ζήτησε το λόγο πριν. Λοιπόν, το πνεύμα του είναι εδώ, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν πειράζει, θα, θα γεμίσω εγώ το κενό και εγώ θέλω να ρωτήσω τον Τζον Βόλτς για την πιθανότητα του εξή. Θα μπορούσατε να φανταστείτε, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων, ε, καινοτόμων προγραμμάτων υψηλού κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα είχαν μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας και που μπορεί και να αποτύχαναν, αλλά και πάλι τα χρήματα αυτά να μην τα ζητήσει πίσω η Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Μπορούμε αυτό να μπορεί να το σκεφτούμε για την ανάλυση του κινδύνου. Γιατί φαντάζομαι περισσότεροι από εσά θα συμφωνείτε μαζί μου ότι η καινοτομία είναι ένα επικίνδυνο τομέα, ιδιαίτερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω σχετίζεται με τα όσα είπε ο κύριος ε, Γέγκερ ε, για αυτά τα προγράμματα, για αυτή την κατηγορία προγραμμάτων, θα, των καινοτόμων προγραμμάτων, θα ήταν υποχρεωτικό να υπάρχουν περισσότεροι από ένας εταίρους, δηλαδή που θα δεν θα απευθύνονταν μόνο σε μία επιχείρηση, σε μία περιφέρεια, αλλά που θα μπορούσαν να, να, να ξεπερνούν τα σύνορα της μιας περιφέρειας. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε προς αυτή την ε, λύση και στην κυρία Κατάνα ε, γιατί είπατε βασικά ότι στη Ρουμανία αντιμετωπίζεται ακόμα την πρόκληση της πολιτιστικής αλλαγής, της αλλαγής νοοτροπίας όσον αφορά την καινοτομία. Πιθανότητα δεν ισχύει αυτό μόνο για τη Ρουμανία, είναι εν γέννη ισχύ στην Ευρώπη. Αλλά μείνουμε στα νέα κρατημέλη, είναι ένα ευρύτερο θέμα, όχι μόνο ε, για τη Ρουμανία. Ε, στο πλαίσιο αυτό λοιπόν πώς βλέπετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε από τη στήριξη σε κάποια μεμονωμένη καινοτόμα ε, επιχείρηση και το δικό της ε, project σε μια στρατηγική προσέγγιση περιφερειακού επίπεδου όπως έγινε στο δυτικό Μπραμπάντ ε, στις κάτω χώρες. Πιστεύετε Πώ μπορεί να γίνει ήδη τώρα, γιατί η προσωπική μου εμπειρία με τι ε, κάτω χώρε είναι ότι άρχισαν ε, με ένα τέτοιο, ε, με μια τεράστια όθηση και τώρα εμείς ακολουθούμε. Οι περισσότερες μάλιστα περιφέρειες έχουν αρχίσει με αυτή την περιφερειακή στρατηγική προσέγγιση. Και επίσης ε, μιλήσατε για ότι δεν χρειάζονται μόνο χρήματα, αλλά και επιπλέον στήριξη, βοήθεια που δεν είναι οικονομικού χαρακτήρα. Ένα είδος ε, ε, παρακολούθησης, στήριξης, προώθησης που μπορεί να συνοδεύει την, σε καινοτομίε. Το προτείνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της καινοτομίας και της χρηματοδότησης της στο μέλλον. ότι δηλαδή θα ήταν μια απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να φτάσουν οι μικρομεσαίες στην ε, χρηματοδότηση. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτούς τους επιπλέον όρους έτσι ώστε η Κομισιόν να μπορεί να βοηθήσει να εντοπίσουμε καταρχήν ποια θα είναι αυτή η επιπλέον ε, ε, χρηματοδότηση θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε ένα τέτοιο είδος, να, να, να θέσουμε ένα τέτοιο όρο, ώστε να μπορεί να υπάρχει και μια συνοδευτική ε, παρακολούθηση. Και αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, νομίζω πως δεν υπάρχουν, θα ήθελα να ζητήσω τα σχόλιά σας ε, από τους συζητητές. Ε, Καταρχήν είπατε για χρήματα για ε, τη Νότιο-Δυτική Ολλανδία. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση και αυτή συμβάλλει. Εγώ δεν σας έδειξα τι χρήματα βάζει η εθνική κυβέρνηση, ποιο ήταν το ποσό που βάζει η εθνική κυβέρνηση στην περιφερειά μας. Έχουμε έξι περιφέρειες και η Ολλανδική κυβέρνηση στη δική μας περιοχή βάζει μόνο 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έχουμε διαρκώς λοιπόν το πρόβλημα πως έχουμε περισσότερα καλά προγράμματα από όσα μπορούμε να στηρίξουμε. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι με την ε, κατασκευή μιας περιφερειακής ατζέντα μπορεί κανείς να διαχειριστεί το πρόβλημα της συγχρηματοδότησης. Άμα βάλει όλα τα χρήματα δηλαδή σε ένα μεγάλο πακέτο λύνει το πρόβλημα. Και ήδη τα περασμένα χρόνια είδαμε ότι υπάρχει αυξανόμενη συνένεση για να κάνουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Η εθνική κυβέρνηση, η Περιφερική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την ίδια ατζέντα. και έτσι ήδη τα καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, θα πρέπει κανείς να αποφασίσει να συστήσει μια ημερήσια διάταξη με μια κυβερνητική δομή που θα στηρίζει την ε, ατζέντα αυτή και ούτω καθεξής. Και φαντάζομαι πως η απάντηση είναι ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν κανείς επιταχύνει την κοινοτομία, πάντα λείπουν τα χρήματα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να έχετε υπόψη το, το εξή, ότι χρειάζονται κάποια χρήματα και το, το ανέφερα ήδη, χρειάζονται κάποια χρήματα για τη διαδικασία, για να ξεκινήσει αυτή η αρχιτεκτονική της συνεργασίας, διότι δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή. Και σας τόνισα ήδη πως είμαστε μία μέση περιφέρεια το τι μπορούμε εμείς να πετύχουμε είναι δυνατόν και στις άλλες περιφέρειες, γιατί δεν έχουμε τεχνικό πανεπιστήμιο, δεν έχουμε την, ε, τα κεντρικά της Φίλιπ στην περιφέρειά μας. Ε, μπορούμε να τα καταφέρουμε όμως αν συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες σε κάποιους τομείς, όχι σε, στα πάντα, Θα ήθελα και εγώ να παρέμβω στις δύο ερωτήσεις που μου απευθύνθηκαν άμεσα και συνδέονται μεταξύ τους. Η ερώτηση για την οικονομική, λογιστική και μηχανική. Δεν έχω υπόψη μου κάποιες αξιολογήσεις ή εκθέσεις προόδου για τον Τζέρεμι, για τον Τζέσικα σε σχέση με την αστική ανάπτυξη. Ε, Αυτά τα προγράμματα ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο, άντε 18 μήνες. Ιδιαίτερα για τον Τζέρεμι, όπου ο βασικός διαχειριστής είναι η EIB, δεν έχουμε ακόμα αξιολόγηση, αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Πόσο, πόσο αποτελεσματικό θα είναι, πόσε σε ε, μικρομεσαίε θα ε, ωφεληθούν, θα πρέπει να επανέλθουμε αργότερα. Δεν έχουμε ακόμα κάποια αξιολόγηση. Αυτό τώρα που νομίζω ότι βρίσκεται και στο site μας είναι ότι κάναμε μια αξιολόγηση αυτών των μέσων ε, στο προηγούμενο πρόγραμμα και δημοσιεύθηκε πριν από 1,5 χρόνο ή 2 χρόνια. Αν θέλετε μπορώ να σας το διαβιβάσω στην Επιτροπή. Είναι μια πιο ad hoc προσέγγιση γιατί δεν είχαμε την πρωτοβουλία Jeremy που είναι πιο δομημένη, πιο κατανοητή, πιο γενική. Δεν τολμώ λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάνω κάποιε προκαταρκτικέ παρατηρήσει για το ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Σίγουρα, βέβαια, η Κομισιόν γνωρίζει την έλλειψη δημόσιου χρήματος και αναζητούμε τρόπους ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για να ελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και άλλους ε, ε, προμηθευτές κεφαλαίου. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, είναι μια λεπτή ισορροπία το να βρούμε τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να λειτουργήσουν όλα αυτά, να είναι αποδοτικά και βεβαίως να επενδύσουν και στις σωστές εταιρείε. Και αυτό με φέρνει στην ερώτηση της Προέδρου. Ότι δηλαδή είναι αυτοπόδεικτο ότι δεν επενδύει κανεί σε μια εταιρεία άμα ξέρει πώ θα αποτύχει. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίσει τις ε, οργανισμού περιφερικής ανάπτυξη, ε, να επενδύουν σε εταιρείε που αν και μπορεί να είναι επικίνδυνε, μπορεί να επιτύχουν και να επιτύχουν πολύ θεαματικά. Και αυτό ακριβώ ε, είναι που διέπει και το κεφάλαιο το επισφαλές. Διότι δηλαδή επενδύει κανεί σε διάφορε εταιρείε που συχνά αναπτύσσονται πολύ γρήγορα αλλά που λειτουργούν σε επικίνδυνου τομεί τομεί και ανέχεσαι ένα επίπεδο αποτυχία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όμω για τον διαχειριστή του χαρτοφυλακίου είναι ότι θα πρέπει να έχει εμπορικά κριτήρια υπόψη του όταν επιλέγει καθέναν από του υποψηφίου. Πρέπει να εξετάσει το, το επιχειρηματικό του πλάνο και γι' αυτό και χρειάζεται του ειδικού ώστε να, μπορεί να, εξετά, να μπορούν να εξετάσουν κάθε περίπτωση χωριστά για τι επενδύσει. Δεν επενδύει κανεί βέβαια άμα ξέρει ότι θα αποτύχει η εταιρεία στην οποία επενδύει, αλλά συχνά οι εταιρείε ε, ρισκάρουν. Δεν βλέπουμε λοιπόν μόνο το ποσοστό επιτυχίας αλλά και το ποσοστό απόδοσης των επιχειρήσεων και σε πιο τεχνικό επίπεδο η Κομισιόν αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των εταιριών που πτωχεύουν σε μια φυσιολογική διαδικασία και αυτό συμπεριλαμβάνει το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης βέβαια όπου οι αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης έχουν λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να ε, εκτιμήσουν σωστά το μέγεθος της ε, ε, επιδότησης, αλλά παρόλα αυτά η επιχείρηση αποτύχει, πτωχεύσει, θα συνεχίσουν παρόλα αυτά να δουν τις επιδοτήσεις. Βέβαια τα κριτήρια, οι όροι από την αρχή είναι πολύ στεναροί. Υπάρχει όμως ένα, μια ανοχή για την αποτυχία και βέβαια ε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους όσο, γίνεται όσο αυτό είναι δυνατόν. Και βεβαίως ε, θα ενημερωνόμαστε καταλήλως. Σας ευχαριστώ. Θα επανέλθω ε, στα αυτά τα δύο θέματα. Είναι σημαντική η συνοδεία, η συνοδευτική βοήθεια. Είναι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας των κοινοτικών κονδυλίων. Να θυμίσω δύο στοιχεία. Στις μελέτες που έχουμε κάνει στο EMPM ε, είναι προφανές ότι εκεί που υπήρξε εταιρική σχέση και παρακολούθηση και συνοδεία προς τις εταιρείες ε, ένα, απορροφήθηκαν σημαντικά διαρθρωτικά κονδύλια τα οποία ωφέλησαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ εκεί που δεν έγινε αυτό δεν μπόρεσαν να ωφεληθούν από τα κοινοτικά κονδύλια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μόνο κάποιες μεγάλες εταιρείε. Έπειτα, μιλήσατε για χρηματοδότηση των επικίνδυνων ε, εταιριών. Αν αυτό συνδεθεί με πολύ καλή παρακολούθηση και συνοδεία, αυτόματα μειώνεται και ο κίνδυνος. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στις δράσεις για την ε, τραπεζική χρηματοδότηση, όπου συνήθως γίνεται αυτό με μια, όλο, όλο και περισσότερο μάλλον γίνεται με την συνοδεία ενδιάμεσων ε, οργανώσεων και οργανώσεων των επιχειρήσεων. Και μάλιστα αυτή είναι και η αρχή της εγγύησης για τις μικρομεσαίες. Οι ταράπες ξέρουν πολύ καλά ότι αν δημιουργηθεί ένα σύστημα που μαζί με την χρηματοδότηση συνοδεύουν με συμβουλές, παρακολούθηση, στήριξη από πλευρά των ενδιάμεσων οργανισμών, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος. Δύο στοιχεία να σας πω σε σχέση με τη σημασία αυτής της συνοδευτικής βοήθειας. Έχουμε πολύ λίγα στοιχεία σε κοινοτικό επίπεδο για τα ωφέλη των εν λόγω ε, επιχειρήσεων από τα διευθυντικά ταμεία. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα που μας δόθηκαν από δύο νέα κρατημέλη τα τρία, για τρία χρόνια. Είναι το παράδειγμα της Πολωνίας και της Τσεχίας. Για κατά τρία χρόνια λοιπόν, τρία έτη, 3.000 μικροεπιχειρήσεις της Πολωνίας και 3.000 μικροεπιχειρήσεις της Τσεχίας ωφελήθηκαν από τα διορθωτικά ταμείο. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά διότι αυτές οι επιχειρήσεις δημιούργησαν χονδρικά πάνω από 9.000 θέσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι χάρη στη συνοδεία 20.000 επένδυση από τα διευθυντικά ταμεία οδηγεί στη δημιουργία τριών νέων θέσεων απασχόλησης ανά εταιρεία. Και όλα αυτά συνδέονται και πάλι της συνοδείας, όπως σας είπα, συνοδευτικής βοήθειας και στήριξης στις εταιρείες. Ναι, Γιάννη μια πολύ σύντομη παρατήρηση στα όσα είπατε. Γιατί με ρωτήσατε ποια είναι η κρίσιμη μάζα για τα διαρθρωτικά ταμεία. Κοιτάξτε, Μήπως έχουμε κάποια ποσοστά εδώ να δώσουμε, γιατί μου είπατε αν έχουμε την ιτορική σχέση, αν είναι η κρίσιμη μάζα διαθέσιμη, μπορείτε κάπως αυτή να την ποσοτικοποιήσετε. Δεν εκφράστηκα καλά ζητώ συγγνώμη. Θα έλεγα πως εάν αυτή τη στιγμή έχουμε την συνοδεία και την ε, συμβουλή των ενδιαμέσων ε, φορέων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν εύκολη πρόσβαση στα διαφορετικά ταμεία. Μόνοι στους όμως, χωρίς συνοδεία, δεν έχουν πρόσβαση, δεδομένου ότι είναι πολύ δύσκολο και οι διαδικασίες και οι προετοιμασίες των φακέλων. Εάν λοιπόν θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα διαφορετικά ταμεία. Ένα από τα κριτήρια τα οποία είναι ουσιαστικά και ζωτικά είναι να περάσουν από ενδιάμεσους φορείς προς μια πολιτική η οποία θα βοηθάει το coaching, την συνοδεία και την ε, βοήθεια. Η κυρία Κατάνα θέλει να πάρει το λόγο. Νομίζω πως θα πρέπει οι περιφέρειες να είναι οι βασικοί παίκτες έτσι ώστε αυτές οι καινοτόμες λύσεις να προκριθούν. Θα πρέπει δηλαδή τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν μια τακτική, μια διαδικασία, μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Και νομίζω πως για το κατά πόσο θα πρέπει να, να συγκεράσουμε όλα τα ποσά, να σας πω πως και τα εθνικά ταμεία και τα κονδύλια και τα κοινοτικά είναι πολύ σημαντικά και καλά να χρησιμοποιούνται μαζί. Ο κ. Γιάγκερ. Εσείς κύριε Γέγερ, το ερώτημα εάν η συγχρηματοδότηση είναι σκόπιμη ή αν ίσως θα ήταν σκοπιμότερο να διατίθεται η πόρη στην ίδια τη χώρα. Για αυτό το θέμα εγώ θεωρώ ότι στα διαρθρωτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπω και μια βάση ώστε να ζητηθεί η συγχρηματοδότηση και στο επίπεδο της περιφέρειας. Γιατί ελάχιστες περιφέρειες διαθέτουν και τους φορείς εκείνους που θα επιτρέψουν τη χρήση των κονδυλίων αυτών. Αν αρχίσει λοιπόν αυτό θα υπάρξει και μια ροή που θα κινητοποιήσει ε, τους ενδιαφερόμενους να ε, προσφέρουν και συγχρηματοδοτήσεις. Εάν δεν υπάρχει το κίνητρο αυτό, εν τέλει δεν θα δραστηριοποιούνται παρά μόνο αυτοί που ήδη δραστηριοποιούνται. Και ήδη μιλήσαμε για αυτό το υπνότον δυναμικό που δεν εντοπίζεται μονάχα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά σε όλα τα επίπεδα και στα επίπεδα των περιφερειακών κυβερνήσεων και στα επίπεδα των ε, ε, επιμελητηρίων, ε, βιομηχανικών και εμπορικών επιμελητηρίων και, υπάρχει, και εκεί υπάρχει ένα υπνό δυναμικό το οποίο πρέπει να αφυπνιστεί. Για τη χρηματοδότηση λοιπόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς για παράδειγμα τα σχέδια επεκτάσεώς μας τα καταφέραμε να τα υλοποιήσουμε μόνο με, τις, με τη χρηματοδότηση του κρατηδίου μας. γιατί η ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν γίνεται στην τάξη του 10% τον χρόνο. Καμιά φορά γίνεται με διπλασιασμό, τριπλασιασμό και δεκαπλασιασμό ακόμα των ε, ε, δυνατοτήτων ικανοτήτων της περισσότερο. Εκεί προσφέρεται η δυνατότητα αυτή, θα έπρεπε να προσφέρεται η δυνατότητα χρηματοδοτησης ή προσφορά εγγύησεων. Μάλιστα σιγά σιγά ε, προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση των εργασιών της ακροάσεώς μας. Νομίζω ότι απηχώ την άποψη όλων των συναδέλφων όταν λέγω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε, καθώς και πηγή εμπνεύσεως για μας και σας ευχαριστώ που φωτίσατε το θέμα από διαφορετικές γωνίες, προσφέροντας έτσι και τις εμπειρίες σας. Ευχαριστώ και για το ε, θέμα αυτό που θέσατε υπόψη μας, ε, του υπνότοντος δυναμικού Μέχρι τώρα μας έλεγε η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το untapped potential, το ε, δυναμικό που δεν έχει αντιληθεί ακόμα, αλλά τώρα θα αρχίσουμε να μιλούμε και για υπνότον δυναμικό. Εγώ βρίσκω ότι αυτό είναι σημαντική εξέλιξη. Και σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε το έργο σας που είναι χρήσιμο και πιστεύω ότι με κοινή προσπάθεια θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε το υπνότον δυναμικό και στην προσεχή περίοδο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και καλό όλους να σας χειροκροτήσουν. Τώρα ε, θα είμαι πραγματικά ε, ιδιαίτερα αυστηρή όποιος δεν συμμετέχει στην, ε, στους ε, συντονιστές να αποχωρήσει αμέσως από την αίθουσα. Αύριο συναντώμεθα στις 9. Και φέρτε και τις κάρτες σας διότι προβλέπετε ψηφοφορία.